Ο, ο πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας αρχίσουμε ευθύς αμέσως. Σας ζητώ συγγνώμη. Ποτέ δεν αργώ, το ξέρετε αυτό. Αλλά, κύριε Έγγελ, ξαναλέω, ποτέ δεν καθυστερώ. Σήμερα υπήρξε εξαίρεση, διότι προτιμούσα να ξεκαθαρίσω κάποια θέματα της επόμενης εβδομάδας που αποδείχθηκαν πολύ περίπλοκα και ευτυχώς νομίζω τα καταφέραμε. Ζητώ συγγνώμη ιδίω από τον ε, κύριο Επίτροπο, ο οποίος ήρθε μάλιστα και 10 λεπτά νωρίτερα. Ζητώ συγγνώμη. Και αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει χρόνο παραπάνω από τις 3 και 30. Άρα, χωρίς να πω περισσότερα λόγια και χωρίς καν εισαγωγή, θα παρακαλέσω τον κύριο Επίτροπο να αρχίσει. Θα πω μόνο να θυμίσω δηλαδή στους συναδέλφους ότι στις 27 Ενάτου δημοσιεύθηκε ανακοίνωση με το θεματολόγιο της μετανάστευσης και βεβαίω τον ε, καλωσορίζω και τον παρακαλώ να, να μας ε, μιλήσει και για το για τον χώρο Σέγγεν. Ε, παρακαλώ κάντε την εισαγωγική σας ομιλία και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις. Αρχίστε κύριε Επιτροπέ. Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητέ Κλοντ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αξιότιμοι ευρωβουλευτές, πρώτα θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω την πιο πρόσφατη ανακοίνωση για το μεταναστευτικό και για το Σέγγεν. Ατυχώς έχουμε μόνο περίπου μία ώρα, λιγότερο από μία ώρα, παρά το σφιχτό μας χρονοδιάγραμμα και και ε, το γεγονός ότι η συζήτηση ε, οργανώθηκε με, σε πολύ σύντομο διάστημα. ευχαριστώ ε, θα ανταλλάξω απόψεις μαζί σας και είμαι και στη διάθεσή σας αν θέλετε να επανέλθω για να εμβαθύνουμε τις συζητήσεις στα σημαντικά αυτά θέματα. Τώρα για το μεταναστευτικό. Έχουμε διανύσει μεγάλο δρόμο, όμως μένουν πολλά πράγματα να γίνουν ακόμη. Το μεταναστευτικό θα μας ακολουθεί για πολλά χρόνια. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Είναι ατυχές ότι χρειάστηκε κρίση για να εγκρίνουμε και να εφαρμόσουμε μέτρα αλληλεγγύης τα οποία πάντοτε στήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως το σημαντικό είναι να προχωρήσουμε με κοινό τρόπο, χέρι με χέρι, στην κατεύθυνση μιας ε, σταθερής, βιώσιμης διαχείρισης του μεταναστευτικού που να ολοκληρώνει και τη στρατηγική μας για το μεταναστευτικό. Η αδίποτε μελλοντική κρίση θα πρέπει να βρει την Ευρώπη καλύτερα προετοιμασμένη και εξοπλισμένη. Λείπουν κάποια σημαντικά στοιχεία ακόμη και αναφέρομαι στην προτινόμενη μεταρρύθμιση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου που ήταν και παραμένει μια από τις προτεραιότητές μας. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, να συνεχίσουμε να σώζουμε ζωές ανθρώπων, να προστατεύουμε τα παιδιά που βρίσκονται σε μεταναστευτικές ροές, να αναπτύσσουμε νόμιμους δρόμους για την έλευσή τους στην Ευρώπη, να προστατεύουμε τα εξωτερικά μας κοινά σύνορα, να καταπολεμούμε τα δίκτυα των παράνομων διακινητών και να επιστρέφουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον προηγούμενο μήνα εγκρίναμε ε, νέο σύνολο προτάσεων για τα υλοποιήσιμα στοιχεία της, ε, ε, του θεματολογίου. Λοιπόν, χρειάζεται μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου, ενίσχυση των νόμιμων οδών, πιο αποτελεσματική πολιτική για τις επιστροφές και την εξωτερική διάσταση, το Partnership Framework for Migration, για την μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου έχει έρθει η ώρα να περάσουμε από την διαχείριση της κρίσεως και τους μηχανισμούς ad hoc σε μια διαρθρωμένη λύση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Ένα μελλοντικό βιώσιμο και προβλέψιμο πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται στην ανάληψη ευθύνης και στην αλληλεγγύη με, να είναι αποτελεσματικό και έντιμο. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή σας θα ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα επί της εκθέσεως της κυρίας Βίξτρομ. Όπως έχω πει κάτι επανάληψη. Ανέμενα ισχυρή εντολή από το Κοινοβούλιο για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στο Συμβούλιο. Εκφράζω λοιπόν τις ευχαριστίες μου και στην εισηγήτρια και στους και εισηγητές όλων των πολιτικών σας ομάδων για τη σκληρή δουλειά, για την στήριξη και για την δέσμευσή τους ε, στο σημαντικό αυτό θέμα. Εφόσον τόσο πολλές πολιτικές ομάδες με μέλη που προέρχονται από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, με διαφορετικές προσεγγίσεις, με διαφορετικές εμπειρίες. Εφόσον όλοι αυτοί κατορθώνουν να συμφωνήσουν για τις προτεραιότητες της αναθεώρησης του Δουβλίνου, ε, θα πρέπει και το Συμβούλιο να μπορέσει να το πράξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ προσωπικά είμαστε διατεθειμένοι και έτοιμοι να παίξουμε τον ρόλο μας, να είμαστε εύκαμπτοι υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχές της ευθύνης και της αλληλεγγύης γίνονται σεβαστέ και ότι καμία χώρα μέρο δεν μένει μόνη τη, δεν την αφήνουμε μόνη τη. Εν τω μεταξύ θα χρειαστεί να συνεχιστεί η πρόοδος και για όλες τις άλλες προτάσεις μεταρρυθμίσεω του συστήματος ασύλου και οι χώρε μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να επιδεικνύουν ελληνική με την Ιταλία και την Ελλάδα. Τώρα, για την επανεγκατάσταση. για την μετεγκατάσταση μάλιστα, θα πρέπει να γίνει ο προτιμόμενος τρόπος για την ε, αποκατάσταση των ε, προσφύγων. Άνθρωποι δηλαδή που χρειάζονται προστασία δεν θα πρέπει να βασίζονται πλέον στην εντό εγών παροχή υπηρεσιών από εγκληματικέ οργανώσει για να φτάσουν να σώσουν τι ζωέ του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και έχουμε κάνει μια πρόταση για ένα ενωσιακό πλαίσιο μετεγκατάσταση τον προηγούμενο Ιούλιο. Γνωρίζω ότι η σχεδιαζόμενη έγκριση τη έκθεση Λίμπε για την πρόταση γίνεται αύριο και ευχαρίστω θα στηρίξω τι διαπραγματεύσει μεταξύ των μερών για να μπορέσει να εγκριθεί σύντομα. Εν τω μεταξύ και μετά τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει έκκληση προς τις ε, χώρες μέλη να μετεγκαταστήσουν τουλάχιστον 50.000 άτομα μέχρι τέλη του Οκτωβρίου 19. Εμείς υποστηρίζουμε την έκκληση αυτή με χρηματοδότηση μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Αναμένουμε από τις χώρες μέλη να αποκριθούν. Έχω κάποια ενθαρρυντικά νέα που θα μπορέσω να επιβεβαιώσω μετά από το Συμβούλιο που θα γίνει την Παρασκευή Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνη. Οι χώρε μέλη, ενθαρρύνουμε τι χώρε μέλη να αναζητήσουν τρόπου να εγκαταστήσουν προγράμματα προσέλκυσης ιδιωτικών ε, ε, δωρητών που θα προσφέρονται από ε, ιδιωτικές ομάδες ή από ομάδες ιδιωτών δηλαδή και έχουμε ζητήσει από την ΆΖΟ να προωθήσει τέτοια προγράμματα με τη συνεργασία ενδιαφερομένων χωρών μελών. Τώρα, για την νόμιμη μετανάστευση. Γνωρίζουμε ότι είμαστε μια ήπειρος που πάσχει από τη γύρανση του πληθυσμού και που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έλλειψη δεξιοτήτων. Πρέπει να ανοίξουμε λοιπόν νόμιμους δρόμους, νόμιμους διάβλους για να προσελκύσουν οι χώρε μετανάστες που έχουν τις αναγκαίε δεξιότητες για να ενισχύσουν το εργατικό δυναμικό. Η οικονομική μετανάστευση δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι παράτυπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη ώστε στο 2018 να συντονίσει πιλωτικά προγράμματα για την νόμιμη μετανάστευση με επιλεγμένες τρίτες χώρες και να προσφέρει χρηματοδότηση στις χώρες εκείνες μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Βεβαίως ε, αυτά εξαρτάται από τις ανάγκες που διαπιστώνουν στις αγορές εργασίας τους. Θα συνεχιστούν και οι διαπραγματεύσεις για την γαλάζια κάρτα. Οι στόχοι μας θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξοι για να προσελκυστούν μετανάστες με υψηλές δεξιότητες και προσόντα. Βασιζόμαστε στην εμπειρία της εισηγήτριας και του πρόεδρου Κλοντ Μωράης, ο οποίος συνεργάζεται με πολύ ε, σημαντικούς εισηγητές, δεν μπορούμε να παραμείνουμε εκεί που βρισκόμαστε, στο status quo. Χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματική πολιτική επιστροφών για να είναι αξιόπιστη η μεταναστευτική μας πολιτική πρέπει να είναι και αποτελεσματική στην επιστροφή προσώπων που δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στις επικράτειέ μας. Αυτό απαιτεί μια σειρά πιο διαρκών προσπαθειών και από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και από την πλευρά των χωρών μελών. Η παρούσα κατάσταση όπου οι περισσότερες από τις μισές αποφάσεις επιστροφών δεν ε, εκτελούνται δεν μπορεί να συνεχιστεί. Στα πλαίσια αυτά, ιδίω ο οργανισμός ακτοφυλακή και συνοριοφυλακής θα πρέπει να παίξει τον συντονιστικό ρόλο για όλες τις προσπάθειες επιστροφών. Με συνδυασμό των προσπαθειών η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ισχυρή, ισχυρότερη δυνατότητα μόχλευσης απέναντι στι τρίτες χώρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επίση έτοιμη να αξιολογήσει εάν ίσως χρειάζονται και πρόσθετα βήματα, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση μιας γνήσιας και αποτελεσματικής ε, προσπάθειας, ενός συστήματος επιστροφών για να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση πιο αποτελεσματικά. Αλλά αυτό δεν αρκεί, διότι χρειάζεται και η προσπάθεια ενίσχυσης των ικανοτήτων των χωρών μελών να διερευνούν το έγκλημα της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Γι' αυτό του χρόνου θα προτείνουμε ένα κοινό πλαίσιο και ξεκάθαρες εντολές για το προσωπικό που αποσπάται σε τρίτες χώρες, για αξιωματούχους συνδέσμους και για να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό του δικτύου των Ευρωπαίων αξιωματούχων σύνδεσης για τη μετανάστευση που έχουν ήδη αποσπαστεί σε 12 χώρες προτεραιότητας για την αντιμετώπιση του εγκλήματος δεν αρκεί χωρίς, ε, αν δεν ασχοληθούμε και με τους παράγοντες που κάνουν ελκυστική την ε, έλευση στην Ευρώπη, τους pull factors. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα διαβουλευτεί με τις χώρες μέλη και με άλλους φορείς για να κατανοήσουν όλοι καλύτερα τον ρόλο που παίζουν οι παράγοντες αυτοί και η ανάγκη να υπάρξουν και αντικίνητρα. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με τοπικές και εθνικές αρχές όσες είναι ε, σημαντικές για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης όπως ε, η κοινωνική ασφάλιση και άλλοι φορείς. Ταυτόχρονα είναι ουσιώδες η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει αλληλεγγύη με την Αφρική. 2,85 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν καταστεί διαθέσιμα έως τώρα από το Ευρωπαϊκό Trust Fund για την Αφρική, για την εξασφάλιση της σταθερότητας και για την αντιμετώπιση των ριζών της παράνομης μετανάστευσης, των αιτιών της παράνομης μετανάστευσης. Με δικαιούχους 26 χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, της λίμνης του Τσάντ και του κέρατος της Αφρικής και της Βόρειας Αφρικής. Το νέο External Investment Plan είναι και αυτό μέρος της δέσμευσης αυτής της Ευρώπης. Αναμένεται να προκαλέσει, να 44 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύσεων σε χώρες εταίρους στην Ασία και αλλού μέχρι το 2030. Χρειάζεται προσπάθεια σε όλα τα μέτωπα και οι χώρες αυτές να δεχθούν την επανεισδοχή παράνομων μεταναστών που προέρχονται από τις χώρες τους. Ρυθμίσεις πρακτικού χαρακτήρα έχουν γίνει ήδη για την επανεισδοχή με ορισμένες χώρες προελεύσεως και άλλες τέτοιες συμφωνίες βρίσκονται στην βάση της διαβούλευσης. Τώρα για το Σέγγεν. Δεν θα επαναλάβω το πόσο σημαντικό είναι το Σέγγεν για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η ενοποίηση. Είναι μια θέση την οποία μοιραζόμαστε όλοι. Έχουμε προτείνει να προσαρμόσουμε ακόμη περισσότερο το σύστημα του Σέγγεν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει απέναντι της Ευρώπη και να είναι ακόμα πιο ισχυρό. Προτείνουμε μια τροποποίηση για τον κώδικα Σέγγεν για την προσωρινή διενέργεια ε, συνοριακών ελέγχων στην περίπτωση που μια χώρα μέλος αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο για την εσωτερική της ασφάλεια ή δημόσια τάξη. Γι' αυτό προτείνουμε από τη μια μεριά τροποποίηση των χρονικών ορίων που προβλέπουν οι ε, ε, τρέχοντες κανόνες και να υφίστανται βέβαια, να υπαχθούν μάλλον και σε αυστηρότερη εποπτεία. Με τα στοιχεία αυτά θέλουμε να εξασφαλίσουμε ώστε οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης να παραμείνουν ένα μέσο ίστατης καταφυγής και οι γειτονικέ χώρες μέλη να συμμετέχουν απολύτως σε μια προσπάθεια να μειώσουν ώστε τον συντομότερο τις αρνητικές συνέπειες επί της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Όταν θα καθίσταται αναγκαίοι τέτοια έλεγχη ταυτόχρονα, υιοθετούμε την πρόταση για την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων για προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι καθώς εκκρεμεί η συζήτηση για τις ε, προτινόμενες ρυθμίσεις, οι τρέχουσες ρυθμίσεις του κώδικα Σέγγεν εφαρμόζονται σωστά. Η σύσταση αυτή μεταφέρει το κοινό μα ε, ενδιαφέρον αλλά και την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών. Θα αρκεστώ σε αυτά τα λόγια αγαπητέ Πρόεδρε, αναμένω να ακούσω τα σχόλια και τις ερωτήσει σας σε αυτή την πρώτη βεβαίως ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Συνάδελφοι, έχουμε αρκετούς που θέλουν να πάρουν το λόγο. Έχουμε μόνο μέχρι τις 3.30 και έχουμε πολύ σοβαρά θέματα και θέματα που τώρα συζητώνται όπως το, το Δουβλίνο. Είναι πολύ ευρύ το ρεπερτόριο, αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι για να μπορέσουμε να ακούσουμε και απαντήσεις από τον Επίτροπο. Ας ξεκινήσουμε με την κυρία Μετζόλα. Ευχαριστώ Κλόντ, ευχαριστώ Επίτροπε για την ε, παρουσίασή σας ε, για την ε, ανακοίνωθεν της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Μετανάστευση και για το ότι ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή μας με ειλικρίνεια στη συζήτηση. Η λειτουργία της ζώνης του Σέγγεν απαραίτητο σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων και να βελτιώνουμε την απόδοσή μας στις επιστροφές και τις επανεισδοχές δεν, δεν μπορεί το ένα να υπάρξει χωρίς το άλλο. Το έχω επαναλάβει αρκούντος, αλλά φαίνεται ότι πρέπει να το ενισχύσουμε αυτό, γιατί τελικά κανένας πολίτης δεν θα έχει εμπιστοσύνη στο Σέγγεν, εάν δεν είναι βέβαιος ότι έχουμε όλα τα, λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα και ότι όλα τα κρατημέλη τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Για τις επιστροφές τις αναφέρατε, αλλά πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε για ένα επιχείρημα για δίκαιη ε, διαχείριση με μετανάστευσης εάν οι επιστροφές ε, παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο. Το 2014 και 2015 μειώθηκε ο αριθμός και εάν αποκλείσουμε και τις επιστροφές στα Δυτικά Βαλκάνια πέφτουμε στο 27%. Ε, αυτό είναι απαράδεκτο και γι' αυτό και η ερώτησή μου είναι ποια θα είναι τα επόμενα σας βήματα ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η πολιτική επιστροφών. Δεύτερον, παρά τι προσπάθειέ μα στην πρόληψη και καταπολέμηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων των διακινητών σε ολόκληρη τη διαδρομή από τι χώρε προέλευση, χώρε διέλευση, καθώ και ε, τα σημεία εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διακίνηση μεταναστών είναι πολύ μεγάλο έσοδο εγκληματικού τύπου. Πρέπει να διακόψουμε αυτή τη διαδικασία που εκμεταλλεύεται τους πιο ευάλωτους. Το 95% των μεταναστών διευκολύνονται από διακινητές και λαθρεμπόρους. Πώς βλέπετε ότι αυτό ε, το ζήτημα θα εξελιχθεί. Οι μελλοντικέ τάσεις περιλαμβάνονται στην τελευταία έκθεση της Interpol, της Interpol και της Europol ε, την περσινή. Τι θα κάνει η Κομισιόν και για τη Λιβύη. Οι Ευρωπαίοι συνοριοφύλακες συνεργάζονται με τους Λίβιους ομολόγους τους και σήμερα ακούσαμε τον κύριο Λετζέρη. Πόσο είμαστε βέβαιοι για τις επιχειρήσεις που γίνονται από τους Λίβιους συνοριοφύλακες και κατά πόσο θα εντοτικοποιηθεί αυτή η συνεργασία στο μέλλον. Ε, τι γίνεται λοιπόν χωρίς τους Λιβίους εταίρους μας για να βελτιώσουμε ε, τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών στη Λιβύη. Ο κύριος Κύρκος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και καλώς ήρθατε Επίτροπε. Θα ήθελα, καθυστέρησα επειδή θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τον Πρόεδρο Μωράζ για την εκδήλωση που έκανε πριν το καλοκαίρι για την κατάσταση στα hot spots στην Ελλάδα με τη κυρία Μακάβαν. Πολύ σημαντικό και μάθαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Και γι' αυτό έχει η πρώτη μου ερώτηση που είναι είδαμε την ύπατη αρμοστία ότι εκφράζει ανησυχίες για τον χειμώνα που έρχεται και θυμόμαστε όλοι τις περσινές φωτογραφίες με τους νεκρούς στη Μόρια. Φαντάζομαι πως συμφωνείτε μαζί μου πως η Κομισιόν πρέπει να κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι της, είτε σαν βοήθεια είτε σαν πίεση, ώστε να μην ξαναδούμε τέτοιες φωτογραφίες που προσβάλλουν τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό. Και η δεύτερη ερώτηση, υπάρχει μια σύγχυση για το καθεστώς των σύρων που έρχονται στα ελληνικά νησιά πριν από το Μάρτιο της ε, συμφωνίας με την Τουρκία, μετά το Μάρτιο της συμφωνίας και αυτό τον καιρό που τελειώνει το πρόγραμμα της με την κατάσταση. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιος εμπίπτει σε ποια κατηγορία. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Coelho, please. Thank you, Chair. I will speak in Portuguese. Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και για τα όσα είπατε σε σχέση με το Σέγγεν ε, θα ήθελα να μιλήσω. Είναι απαραίτητο να επανέλθουμε στο Σέγγεν. Back to Σέγγεν έχουμε πει πολλές φορές και οι προτάσεις που υποβάλλει η Κομισιόν ε, κινούνται προς σωστή κατεύθυνση. Επίσης χαίρομαι για την ατζέντα για τη μετανάστευση γιατί αντιπροσωπεύει μια μεγάλη προσπάθεια από πλευρά τη Ένωση για να διαχειριστεί καλύτερα την ροή μεταναστών και ε, προσφύγων. Όμω ξεκινά από μια προπόθεση στην οποία αναφερθήκατε στην εισήγησή σα ότι δεν είναι τόσο προφανής ότι δηλαδή θα είμαστε εμείς σε θέση να δώσουμε μια αλληλέγγυη απάντηση. Εδώ και εμείς το έχουμε επαναλάβει συχνά, αλλά όπως είπατε επίτροπε ακόμα πρέπει πολλά να γίνουν. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλές διαρθρωτικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί, όμως ισχύει επίσης ότι έχουμε την αίσθηση πως όλα προχωρούν πάρα πολύ αργά. Ένα παράδειγμα, το νέο, ο νέος οργανισμός για το άσυλο που παρά την ε, πολιτική συμφωνία δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί και πολύ συχνά προχωράμε με ad hoc βήματα, αλλά φρύνονται κάπως τα προβλήματα, αλλά δεν λύνονται. Ας πούμε η επανεγκατάσταση, η μεταγκατάσταση μάλλον ε, λίγων χιλιάδων ανθρώπων είναι ένα παράδειγμα αυτού του γεγονότος. Όλα αυτά είναι πολύ επιβαρυντικά για την υλοποίηση της ατζέντα για την μετανάστευση. Βλέπουμε για την Αφρική, βλέπουμε για την μεταγκατάσταση, βλέπουμε ότι το Συμβούλιο γρήγορα αποφάσισε για έναν οργανισμό για τα σύνορα, ενώ ε, σιγά σιγά συζητά και το Δουβλίνο, σιγά σιγά όμω και φαίνεται να ισχύουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανάλογα με το κάθε μέτρο. Οι προτάσει, σα λοιπόν επίτροπε προχωρούν στη σωστή κατεύθυνση κατά τη γνώμη μου, αλλά για εμά, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών από το Κοινοβούλιο, δεν φαίνεται να ακολουθούν τα κράτη-μέλη την ίδια γραμμή. Και αυτό μα ανησυχεί για το Συμβούλιο είναι συνομοθέτης. Η κυρία Έλλη Σλάινα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ Επίτροπε για την ε, ε, συνηθισμένη σας διαθεσιμότητα και για τι πληροφορίε που μα δώσετε σήμερα σε σχέση με το ανακοινωθέν. Εργαζόμαστε σκληρά για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. όπω γνωρίζετε η ομάδα μα εδώ και καιρό έχει δεσμευθεί για να εφαρμοστούν τα όσα απαιτούνται από τι συνθήκε όταν ζητούν αλληλεγγύη και κοινή ευθύνη, μοιρασιά τη ευθύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως ε, επανειλημμένα έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο μα και μέσω τη έκθεση τη κυρία Μπετζόλα και Κέγκε τον περασμένο Απρίλιο. Ήδη έχει χαθεί χρόνο και είμαι, ε, έχω εμπιστοσύνη και εύχομαι ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα μπορέσει να δώσει μια ισχυρή και φιλόδοξη θέση για το Δουβλίνο, να στείλει όντω ένα μήνυμα προς το Συμβούλιο και να δώσει ένα τρόπο στην Κομισιόν ώστε να ξεκινήσει και πάλι και να επιμένει ε, προς το Συμβούλιο για την αρχική της πρόταση που, που, που θα πρέπει να μείνουν κάποια σταθερά στοιχεία. Δηλαδή μεταξύ αυτών είναι σίγουρα και η ανάγκη για κοινέ ευθύνε με έναν μόνιμο μηχανισμό ισότιμο για τις, ε, τη μοιρασιά των ευθυνών και μια πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου δικαίωσε την πρόταση της Επιτροπής για τις μετεγκαταστάσεις όπου βλέπουμε να επικρατεί μια ντροπιαστική διστακτικότητα από πλευρά των κρατών μελών να προχωρήσουν. Απίστευτο ενώ σε τέσσερις μήνες ο Καναδάς το 2016 επανεγκατέστησε άμεσα στην επικράτειά του 40.000 κόσμο, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που δεσμεύτηκαν να μετακαταστήσουν 160.000 κόσμο μέσα σε δύο χρόνια το Σεπτέμβριο του 2015 δεν κατάφεραν αυτό στους 28.000 μετακαταστάσεις. Πραγματικά λοιπόν εγώ σας καλώ από τη στιγμή που θα έχουμε εγκρίνει την ισχυρή και φιλόδοξη μας θέση να ξαναρχίσετε να επιμένετε γιατί το πραγματικό συμβούλιο το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι το κονσίλιο. Εθνικοί εγωισμοί που επικρατούν στο Συμβούλιο ακόμη. Θα ήθελα πραγματικά να κάνω μια ανέκκληση προς την Επιτροπή και να μην μακρηγορήσω άλλο, ώστε να ξαναβρει το πνεύμα της πρώτης ατζέντα για τη μετανάστευση και να μην αφήσει να κάνει πίσω σε αυτές τις τάσεις εξωτερικοποίησης, εξωτερήκευσης των συνόρων μας που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Η κατάσταση στη Λιβύη δεν, με ανησυχεί όχι μόνο εμένα και όλους όσοι είμαστε εδώ, αλλά και την είπα το αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πρόσφατη έκθεση. Μάλιστα και το Συμβούλιο της Ευρώπης ζήτησε διευκρινήσεις από την Ιταλική κυβέρνηση για το ποιε είναι ακριβώς οι συμφωνίες που έχουν συναυθεί με τη Λιβύη, που από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με δημοσιογραφικές έρευνες ε, ενέπλεξαν και τις πολιταφυλακές που πριν διαχειρίζονταν την διακίνηση ανθρώπων. Έχει γίνει μια ε, ε, λογική αντιστροφή στην ε, Λιβύη, γιατί Παλιότερα ζητούσαμε εξασφάλιση καλύτερων συνδικών διαβίωσης των, ε, των ε, προσφύγων, όπου βλέπουμε απάνθρωπες συνθήκε να, να, επικρατούν. Πρώτα πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι αυτοί θα ζουν σε ε, ανθρώπινε αξιοπρεπεί συνθήκε και μετά να κάνουμε συμφωνίε που αφορούν και που, μάλλον, που αναθέτουν στην Λιβική ακτοφυλακή να ασχολείται με αυτού του ανθρώπου. Έχει γίνει μια λογική αντιστροφή λοιπόν που δυστυχώ έχει φρικτά αποτελέσματα μας δείχνουν σε αυτές εικόνες. Μάλιστα. Παρακαλώ, συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος, δύο λεπτά μάξιμου. γιατί τελείως δεν θα έχουμε χρόνο. Χωρισμάνοβα. Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω Επίτροπε, για την ομιλία σας είπατε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες βιώσιμες προσπάθειες ώστε να ε, ε, η, επιστροφή, η πολιτική επιστροφών μας να καταστεί πιο αποτελεσματική. Όμως σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσά, το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό, 36% μόλις για ε, την περίοδο 2014-2015, 1,5 εκατομμύρια ακόμα πρέπει να επιστραφούν, αλλά ε, δεν έχουν επιστραφεί. Επίσης ακούσαμε από τον οργανισμό, τον Ευρωπαϊκό μάλλον οργανισμό ε, για τα σύνορα, ε, ότι θα φτιαχτεί, αλλά ακόμα δεν έχει ε, ξεκινήσει τίποτα. Οπότε διαρωτώμεθα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία και ποιες θα πρέπει να είναι οι νέες εταιρικές μας σχέσεις, σχέσεις με τις χώρες προέλευσης. Ο κύριος Γιούνκερ είπε στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ότι θα πρέπει να επιτείνουμε τις προσπάθειές μας. Δεν θέλω να γνωρίζω εσείς πώς βλέπετε την πρόοδο των επιστροφών των, παράνομα, των παράνομων μεταναστών. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες εσείς περιγράψατε κάποια από τα μέτρα που σκοπεύετε να εφαρμόσετε, αλλά πιστεύετε πως θα αρκέσουν. Ευχαριστώ, κύριο Σέγγελ. Thanks, Claude. Um, Ευχαριστώ, Κλοντ. Εγώ θα ξεκινήσω με το Σέγγεν. Πρέπει να πω πως είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένο σε σχέση με τα όσα μας είπατε και τα όσα μας προτείνετε για τον απλό λόγο ότι δεν βλέπω τα κράτη να θέλουν να εγκαταλείψουν αυτούς τους ανόητους συνοριακούς ελέγχους που έχουν ξεκινήσει ε, γενικώ και ορίστως. Είναι δίθεν έλεγχοι και όλοι το ξέρουμε. Ούτε οι μετανάστες θα πιάσουν, ούτε οι Ρωμακράτες θα πιάσουν με αυτούς τους ελέγχους. Ωστόσο, παριστάνουν ότι κάτι, έχουν να, ότι κάτι κάνουν στους ψηφοφόρους τους. Οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε πάρα πολύ αυστηρός. Εάν προχωρήσετε σε αυτό το νέο προτινόμενο σύστημα σε σχέση με τους όρους που το συνοδεύουν εκτός και αν οι απειλές είναι πολύ συγκεκριμένες και επαληθευμένες θα πρέπει να εγκαταλειφθούν αυτά τα μέτρα όπως θα πρέπει να εγκαταλειφθούν και ένα σωρό άλλα μέτρα όπως ας πούμε το, η κατάσταση επίγουσας ανάγκης ε, που υποτίθεται ότι ισχύει για τη στήριξη στην Αφρική. Εγώ μόλις επέστρεψα από μία συνάντηση με τον ε, πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης. Η Ευρώπη θα πρέπει να συνεννοηθεί για να καταλάβουμε και εμείς από πού μπορούμε να ε, βρούμε κάποια χρήματα μέσα από τα εκατοντάδες προγράμματα που έχει. Ακόμα και με το καταπίστευμα μάλλον με το Ταμείο Εξωτερικών Επενδύσεων που δεν είναι το καταπίστευμα ούτε τα άλλα σχέδια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2016 οι Κινέζοι 40 δις επένδυσαν στην Αφρική, μόνο το 2016. Ακόμα και αν σε 3-4 χρόνια ε, λέγαμε ότι θα επενδύσουμε αυτό το ποσό, η Αφρική δεν το περιμένει αυτό και δεν θα εκριζωθούν τα αίτια των όσων συμβαίνουν. Και τέλος, για τις νόμιμους ε, διάβλους. Ε, Όσο περισσότερο μιλάμε γι' αυτό, τόσο περισσότερο η Ουγγαρία θα, θα μας λέει πως αυτό είναι ε, απαράδεκτο. Και αυτή τη στιγμή ε, ένα σωρό σλόγγαν τέτοιου τύπου κυκλοφορούν, αλλά αυτό πρέπει να γίνει. Είναι αυτό το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, γιατί αν δεν το κάνουμε τότε η πίεση αυτών που διευκολύνουν την παράνομη μετανάστευση δεν θα ε, δώσει καρπούς. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη. Ευχαριστώ κύριε Βραμόπουλε για την εισήγησή σας. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την επιστολή που έστειλε ο Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα του, του Δικαστηρίου του Στρασβούργου στον Υπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας. Θα μπορούσε να τη στείλει την ίδια επιστολή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλες οι Ιταλικές πολιτικές σε αυτό το πεδίο έχουν εγκριθεί από την Ένωση. Και ο Γιούγκερ επένεσε όλος ιδιαίτερος την Ιταλική κυβέρνηση η επιστολή αναφέρει την απόφαση του 2012 ενάντια στην ελληνική πολιτική επαναπατρισμών προς τη Λιβύη και υπογραμμίζει τέσσερα πολύ σοβαρά στοιχεία. Πρώτον, η κατάσταση στην Λιβύη δεν είναι λιγότερο επικίνδυνη από το 2012. Οι επαναπατριζόμενοι κινδυνεύουν να βασανιστούν και να τους δεχτούν απάνθρωποι και υποβαθμιστική συμπεριφορά σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεύτερον, το γεγονός ότι ε, ε, ε, το, μάλλον το γεγονός ότι συμβαίνουν έρευνες και διασώσεις στα ελληνικά ύδατα δεν απαλλάσσει την Ιταλία από την ευθύνη να κάνει τέτοιες επιχειρήσεις διάσωσης. Έπειτα οι άνθρωποι που διασώζονται δεν επιστρέφονται σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος για τη Λιβύη ε, και έπειτα για τη συμπεριφορά των ΜΚΟ η επιστολή ζητά να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων των ΜΚΟ να εξασφαλίζονται και να γίνονται μέσα σε συνθήκες μέγιστης ασφάλειας. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται γιατί στην ουσία οι ΜΚΟ έχουν φύγει από την Κεντρική Μεσόγειο. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητάνε από την Ιταλία αλλά όπως έλεγα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σεσίλ Σας ευχαριστώ, Κλοντ. Ευχαριστώ και εγώ τον Επίτροπο που μας έκανε αυτή την ανακοίνωση, αλλά και την εργασία που καθημερινά εκτελεί στο πλευρό μας. Εγώ ξεκινώ κάνοντας μια παράθεση. Γνωρίζουμε πως το Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει τον Απρίλιο του 2016 το ψήφισμα ε, Κέγγε Μετζόλα με μια γενική προσέγγιση με συγκεκριμένα σημεία που με δυσκολία όμως ε, εφαρμόζονται στην πράξη, ε, γιατί λόγω του εγωισμού των κατών μελών γίνεται δύσκολο να εφαρμοστούν κάποια από τα σημαντικά σημεία που θα πρέπει να μας βοηθήσουν να φτάσουμε σε καλή διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου. Ένα σημείο πολύ βασικό είναι οι νόμιμες οδοί για την μπλε κάρτα έχουμε δουλέψει μόνο, αλλά πρέπει σήμερα να επιμείνουμε ε, για αυτό το δρόμο, γιατί ο κόσμος πάντοτε διαφορετικά θα εμπιστεύεται το λάθος άτομα. Για το Δουβλίνο, για να φτάσουμε στο Δουβλίνο πρέπει πολλά κράτη να εγκαταλείψουν λίγο από τον εγωισμό τους, που τους σωθεί να κλείνουν τα σύνορά τους και να αφήνουν τις ευθύνε στις πλάτες των πρώτων χωρών ε, ε, άφηξης. Να φτάσουμε λοιπόν σε μια καλή συμβιβαστική. Ε, αν πιστεύω, εάν ε, αυτό εδώ το κοινοβούλιο μπόρεσε να δουλέψει και να βρει κοινό, κοινό δρόμο, θα μπορούσε να το καταφέρει και το Συμβούλιο. Η καταπολέμηση του εμπορίου ανθρώπων, ε, το να φεύγουν οι άνθρωποι από τη Λιβύη, εγώ ε, εκτίμησα πολύ το ανακοινωθέν που λέει για ενίσχυση ανθρω... της προστασίας των ανθρώπων που βρίσκονται στη Λιβύη, γιατί ξέρουμε πω η Λιβύη δεν είναι σίγουρη χώρα και να μπορέσουμε να, να πάρουμε τον κόσμο από εκεί όσο γίνεται περισσότερους και να έχουμε μια σαφή εντολή, μια σαφή αποστολή, ιδιαίτερα για τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι άνθρωποι και πρέπει να παρέμβουμε για τα βαθύτερα αίτια αλλά και για να φέρουμε την, την ακουστή φωνή αυτού του κοινοβουλίου. Κάναμε μια, μια γνωμοδότηση που ψηφίστηκε πριν από λίγε μέρες και θα το πάμε αυτό στο summit στην διάσκεψη κορυφής του Αμπιτζάν. Θα είναι η φωνή του Κοινοβουλίου για μια καλή συνεργασία, μια κοινή στρατηγική με τις χώρες της Αφρικής όπου προτεραιότητα είναι οι νέοι και η ανάπτυξη. Κλείνω με δύο λόγια για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Είπατε κάτι πολύ ωραίο, ότι η μεταρρύθμιση του Δουβλίνου αποτελεί τον κρίκο που λείπει για ένα κοινό σύστημα ασύλου. Α κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν ώστε να σταθούμε στο ύψο αυτού του Κοινοβουλίου και τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Μποντίλ Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ. Το σημαντικό είναι να συζητήσουμε το πως οι διάφορες χώρες πρόκειται να τηρήσουν τα υπεσχημένα πως δεν θα κλείνουν τα σύνορά τους και να στέλνουν πίσω τους ε, πρόσφυγες έχουμε ένα 1,3 ε, εκατομμύρια που φύγουν στον Λίβανο μόνο. Ένα στου τέσσερι βρίσκονται στην χώρα. Η Τουρκία έχει πάνω από 3 εκατομμύρια κλπ. κλπ και βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το 2016 έχουμε δώσει ε, προστασία ε, σε 70.000 συντούς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε 400.000 στην Γερμανία που έχουν πάει. Για κοιτάξτε όμως ε, την αναλογία κατά κεφαλή, είναι η Σουηδία είναι εδώ ο πρωταθλητής. Έχουμε 700 πρόσφυγες ανά χιλίους ε, κατοίκους και 10 είναι το αντίστοιχο νούμερο για την Πολωνία. Επομένως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει κάποια προσπάθεια. Περιμένουμε με περιέργεια να δούμε κύριε Επίτροπε πώς θα μπορέσετε να πείσετε όλες τις χώρες να τηρήσουν τις ε, υποχρεώσεις τους πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις διαδρομές της νόμιμης μετανάστευσης. Έχουμε την οδηγία για την μπλε κάρτα, αλλά καλύπτει μόνο αυτούς που έχουν ε, ιδιαίτερες δεξιότητες. Πάρα πολλοί πρόσφυγες εμφανίζονται ε, ως τέτοιοι και στην ουσία είναι οικονομικοί μετανάστες. Το θέμα είναι το να μην προσπαθούμε να τους ε, διώξουμε το γρηγορότερο. Θα πρέπει να μπορούν να εμφανιστούν και με νόμιμο τρόπο στην Ευρώπη. Επίτροπε, ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την ε, αναλυτική ε, εξιστόρηση των δράσεων στις οποίες κάνει η Επιτροπή και εσείς προσωπικά. Ήθελα να σας ρωτήσω, ε, σε σχέση με τη χώρα μου την Ελλάδα, ξέρουμε ότι 26 Σεπτεμβρίου τελείωσε το πρόγραμμα αυτό της μετεγκατάστασης, λειτουργήσε σε κάποιο βαθμό ικανοποιητικό, φυσικά υπάρχουν προβλήματα. Τελευταία, βλέπετε, πληροφορήστε κι εσείς ότι έχουν αυξηθεί οι ροές παρά το γεγονός ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας λειτουργεί και σίγουρα πετράπει το χειρότερο, όμως έχει αρχίσει και υπάρχει μια ε, αύξηση των ροών ε, προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας. Ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, ή τι έχετε σκεφτεί σαν μια διάδοχη κατάσταση της μετεγκατάστασης μετά τη λήξη της 26 Σεπτεμβρίου, αν υπάρχει δηλαδή μια διάδοχη κατάσταση, με το δεδομένο ότι χτες ο, υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, Έλληνη υπουργός, εξήγηλε την σύσταση και δημιουργεί ακόμη πέντε νέων ε, κέντρων ε, εξέτασης και φύλαξης των ανθρώπων αυτών, νοουμένου ότι λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες ροές. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ορισμένες από αυτές έχουν κάποια επικάλυψη μία με την άλλη. Αλλά θα απαντήσω όσο είναι δυνατόν. Η κυρία Μέτσολα στην αρχή. Είπε ότι θα πρέπει να έχουμε μια σφαιρική στρατηγική και συμφωνώ μαζί της. Αυτό το λέμε ευθύς εξ αρχής. Επίσης, πρόκειται σε τακτά διαστήματα να σας αναφέρουμε την σημειωθήσα πρόοδο. Και θέλουμε να εξασφαλίσουμε το ότι τα σύνορα της ε, Ευρώπης αλλά και τα θαλάσσια σύνορα φυλάσσονται και επίσης θέλουμε τα κράτη-μέλη να αξιοποιούν τις ε, δυνατότητές μας όσο γίνεται περισσότερο. Απαντήσω ελληνικά στον κύριο Κύρκο, μια με ρωτήσατε στα ελληνικά. Να σας πω ότι συμφωνώ με την παρατηρήση σας. Εικόνες σαν και αυτές που ζήσαμε τον προηγούμενο χρόνο δεν πρέπει να επαναληφθούν. Κατά τη διάρκεια των ε, επίσημων επαφών που είχα στην Αθήνα με την ηγεσία της χώρας και με τους αρμόδιους υπουργούς ε, δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε οι συνθήκες στα νησιά, ακόμα και στην περίπτωση που επιδεινωθεί ο καιρός, ε, να είναι ανθρώπινες και τόνισα ότι και εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, θα συνεχίσει να προσφέρει τη δική της ε, βοήθεια. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το ξαναζήσουμε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ε, ερώτησης που υποβάλλατε, <clears throat> οι αποφάσεις για τις ε, μετεγκαταστάσεις αφορούν σε εκείνους που ζητούν άσυλο και που προέρχονται με μέσο ευρωπαϊκό όρο αναγνώρισης πάνω από 75%. Η θέση των κρατών μελών ήταν σαφής ότι δεν θα μετεγκαταστούσαν εκείνους που έφτασαν στα νησιά, που αφήχθησαν στα νησιά μετά την θέση σε εφαρμογή της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Οι μετανάστες που έφτασαν στα ελληνικά νησιά μετά την 20η Μαρτίου του 2016 εμπίπτουν ακριβώς στο πεδίο εφαρμογής της ε, δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η δε πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα νομιμοποιείται να κηρύξει ως απαράδεκτες τις δύο υποεξέταση υποθέσεις σύρων καθώς και να προχωρήσει στην επιστροφή τους στην Τουρκία στην βάση ότι η Τουρκία αποτελεί ασφαλή τρίτη χώρα. Η Ελλάδα πρέπει πλέον να επιταχύνει την ε, εφαρμογή αυτής της δήλωσης εξετάζοντας βέβαια κάθε περίπτωση ξεχωριστά και σεβόμενη όλες τις απαραίτητες εγγύησεις. Η ταχεία και διαρκής εφαρμογή της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας θα συμβάλλει στην μείωση των αριθμών όσων συνεχίζουν να φτάνουν παράτυπα στα ευρωπαϊκά σύνορα. Παράλληλα, όπως γνωρίζετε, ενισχύουμε κατά προτεραιότητα τους νόμιμους ε, διάβλους και αναμένω ότι τα κράτη-μέλη θα προχωρήσουν σε νέες δεσμεύσεις για τις μετεγκαταστάσεις. Αυτό είναι σημαντικό όπως αντιλαμβάνεστε καθώς θα δώσει τη δυνατότητα σε σύρους που βρίσκονται όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και σε άλλες γειτονικές χώρες όπως ο Λίβανος και η Ορδανία να ακολουθήσουν νόμιμες οδούς για να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να καταβάλουν χρήματα σε εγκληματικές οργανώσεις και στους διακινητές και βέβαια το σημαντικότερο να εκθέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Uh, uh, Yes. All... Ναι, έχετε δίκιο. Όλα τα στοιχεία της αναθεώρησης του κοινού σύστηματος ασύλου θα πρέπει να ολοκληρωθούν, θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε περισσότερο και αυτό και κάνουμε και σας επαναλαμβάνω ότι προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση και αναθεώρηση του συστήματος. Και γι' αυτό και χέρι-χέρι με την Αστωνική Προεδρία προσπαθούμε να βρούμε μια συμβαστική λύση αποδεκτή από τα κρατή μέλη, ούτως ώστε να υπάρξουν εγγύσεις ότι δεν θα μείνει μόνο τις προσπαθειές του κανένα κρατός μέλος ε, μέσα στην κρίση του μεταναστευτικού και πάρα πολλά από τα θέματα που πρέπει να ρυθμίσουμε είναι αλληλοσυνδεόμενα και φυσικά συνδέονται όλα με τον κανονισμό του Δουβλίνου. Οπότε πρόκειται να εγκριθεί αυτή η έκθεση, όπως λέγαμε, η έκθεση του την επόμενη εβδομάδα. Και αν έχετε εσείς μια ισχυρή εντολή, αυτό θα είναι ισχυρό μήνυμα και προς το Συμβούλιο. Τώρα όσον αυτό που είπε η κυρία Σλάιν, συμφωνώ και υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση του Συμβουλίου ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου του 2017 και η υποχρέωση κατάσταση ισχύει για όλους όσους έχουν δικαίωμα προ τούτο. Στην Ιταλία, την Ελλάδα, πριν αυτήν την ημερομηνία. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν την ε, υλοποίηση μετά τις 26 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι το να αφήσουμε μόνες τους την Ιταλία και την Ελλάδα που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Αλλά για να δούμε και την ε, άλλη όψη, την θετική όψη. Θα πρέπει να μην σκεφτούμε, να μην, να μην ξεχάσουμε ότι όσο αφορά τις έχουμε επιτυχία κατά 90% χάρη στη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών των κρατών μελών και των διεθνών μας εταίρων έχουμε με την καταστήση πάνω από 30.000 ή 2.200 μηνιαία. Οπότε με την εφαρμογή του συστήματος που θεσπίστηκε δημιουργήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνη και έτσι μπορέσαμε να διαχειριστούμε την κρίση. Πολύ που βάλατε σε σχέση με την ε, Λιβύη. Οι συνεχείς μας προσπάθειες είναι να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε στην αποστολή μας εκεί, να βοηθήσουμε το, την υπηρεσία του ΟΗΕ και να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα και για αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό η υπηρεσία του IOM, των ε, μετανάστευση αλλά και η αρμοστία του ΟΗΕ θα πρέπει να βοηθούν και σε επίπεδο ασφάλειας. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό οι λιβικές αρχές να συνεργαστούν περισσότερο με αυτές τις ε, οργανώσεις. Θα πρέπει να εγγυηθούν την ασφάλεια του προσωπικού. Θα πρέπει να δοθεί στο προσωπικό αυτών των ε, οργανισμών ε, ελεύθερη πρόσβαση όπου χρειάζεται να κάνουν τη δουλειά τους θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις σχετικές συστάσεις. Επίσης έχουμε χρηματοδοτήσει με 46 εκατομμύρια την ε, Ιταλία για το δικό της πρόγραμμα. Έτσι πιστεύουμε ότι θα βοηθηθεί η Λιβύη και σιγά σιγά θα μπορέσουν να ελέγξουν τα νότια σύνορα της χώρας. Τώρα είμαστε σε συνομιλίες με τις Ιταλικές Αρχές για κάποιο είδου εξεταστική επιτροπή, ούτως ώστε μόλις υπάρχουν οι κατάλληλες συνέχειες ασφαλείας να γύρει αυτή η αποστολή και στο μεταξύ προσπαθούμε να αξιολογήσουμε το πώς θα έχουμε κάποιο είδου ε, πρόληψη και να υπάρξει καλύτερος έλεγχος στα νότια σύνορα της Λιβύης ούτως ώστε να εντείνουμε τις δικές μας παρεμβάσεις. Και η κατάσταση ξέρουμε ότι είναι δύσκολη, οπότε προσφέρουμε με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης βοήθεια. Βοήθεια ούτως ώστε να υπάρξει εκούσια επιστροφή όσο γίνεται περισσότερων οικονομικών μεταναστών που έχουν παγιδευτεί στην Λιβύη. Οπότε αυτό το πρόγραμμα χέρι-χέρι με την υποκερμοστή το Θα ξεκινήσει αυτό τον ε, μήνα και θα γίνει και κάποιο είδους κατεπίγουσα ε, εκένωση προς ε, τον Νίγηρα. Όσο γίνεται περισσότερων μεταναστών που θα κριθεί ότι χρειάζονται διεθνή προστασία. Φρανκ. Αυτό αφορά και τη δική σου ερώτηση και ο Ρομπέρτα απήντησε και στη δική σου. Είμαι σίγουρη ότι άκουσες ακόμα και αν δεν ήσουν στην αίθουσα. Αυτό το οποίο είπε είναι η εικόνα που έχουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι όσον αφορά τον έλεγχο στα εσωτερικά μας σύνορα. Κάποιοι προβληματίζονται όσον αφορά τι προκλήσει σχετικέ με την ασφάλεια. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανησυχία του. Προσπαθήσαμε εμεί να εξισορροπήσουμε τη μία πρόκληση με την άλλη. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Με την σημερινή μας πρόταση θέλουμε να εξασφαλίσουμε το ότι η... να είναι μόνο τελευταία λύση η αλήθεια των εσωτερικών σύνορων και τα γειτονιάζοντα κράτη-μέλη να περιορίζουν όσο γίνεται λιγότερο την ε, ελευθερία διακίνησης κίνησης ε, και οι έλεγχοι αυτοί να γίνονται μόνο όποτε χρειάζεται. Οι σχέσεις μας με την Αφρική μιλήσαμε σε σχέση με την, κατάσταση και την νόμιμη μετανάστευση. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να προχωρήσουμε να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση στο θέμα μετανάστευση ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αντί των ε, παρανόμων ρορ να έχουμε νόμιμους διάβλους. Οπότε χρειάζεται συνεργασία με τις τρίτες χώρες. αυτό είναι όλο ένα και πιο σημαντικό για τις συνεργασίες με τις χώρες αυτές ούτως ώστε να υπάρξει τέτοια διαχείριση του μεταναστευτικού. Οπότε και έχουμε προτείνει σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και σεβασμός στις εθνικές αρμοδιότητες αλλά και στις ανάγκες της οικονομίας της κάθε χώρας λέγω να έχουμε επομένως κάποιους πιλωτικά προγράμματα για την νόμιμη μετανάστευση με επιλεγμένες τρίτες χώρες ούτως ώστε να βοηθηθούν με ενωσιακή χρηματοδότηση. Φαντάζομαι ότι τα ακούσατε αυτά από τις επαφές σας με τους ε, ε, Αφρικανούς. Τώρα προσπαθούμε να διερευνήσουμε το τι μπορεί να γίνει σε σχέση με αυτό με τις χώρες μέλη. Και για την μετεγκατάσταση, όπως είπα και στην εισήγησή μου, είναι και αυτό θέμα πολύ σημαντικό. Οι γεωγραφικές προτεραιότητες για το πρόγραμμα δράσης και τα μέτρα για βοήθεια προς την Ελλάδα θα φέρει μείωση των πιέσεων στον κεντρικό διάβολο της Μεσογείου. Θα έχουμε περισσότερη ελεγγύη και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σχέδιο ε, του ΟΗΕ της υπάτης αρμοστίας ούτως ώστε να υπάρξει η κένωση των ε, πιο ευάλωτων ε, από την Λιβύη με την κατάσταση από χώρες επίσης, όπως το Τσάδ και την, τον Νίγηρα. Η συνεργασία μας με τον Νίγηρα θα συνεχίσουμε, πάμε καλά, έχουμε κάποια προβλήματα με το Τσάδ και έτσι θα διαχειριστούμε τους εταίρους μας από κοινού τις μεταναστευτικές ροές. Επανέρχομαι τώρα στα ελληνικά, γιατί η κυρία μου υπέβαλε μια ερώτηση. Να λάβω και μια ακόμα φορά ότι η προτεραιότητά μας είναι να μετεγκατασταθούν όσοι είναι επιλέξιμοι στα πλαίσια των δύο αποφάσεων. Παρ' όλα αυτά, τονίζω ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Ιταλία θα αφαιθούν μόνες. Από την πρώτη και όλα στιγμή στηρίζουμε, βοηθούμε αυτές τις δύο χώρες που δέχονται την μεγαλύτερη πίεση και θα συνεχίσουμε. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει και επιχειρησιακά αλλά και οικονομικά τις μετεγκαταστάσεις. Μάλιστα θα συνεχίζουμε να κάνουμε και τακτικές εκθέσεις πρόοδου. Και μπορώ να να σας πω ότι έχω θετικά μηνύματα από πάρα πολλά κράτη-μέλη. Ε, Για την κυρία Κέγκε. Για την δική σας ερώτηση. Πιστέψτε με, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας όσον αφορά ε, τα προβλήματα των μεταναστών. Είναι και δικές μας, οι δικές τους ανησυχίες. Όπου και αν βρίσκονται εκείνοι. Διότι στην ε, Λιβύη, όπως είπα προηγουμένως, ε, είναι θέμα προτεραιότητος. Οι εταίροι μας έχουν αναπτύξει τους σχετικούς ανθρώπινους σπόρους, οπότε και οι οικονομικοί μετανάστες που το επιθυμούν να μπορούν να γυρίσουν στη χώρα τους. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας σε αυτό το μέτωπο αυτό. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Και Ελπίζω ότι θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα. Νομίζω ότι απήντησα σε όλες τις ε, ερωτήσεις. Δεν ξέρω, Πρόεδρε, τι άλλο θέλετε από μένα, αλλά όποτε θέλετε να ξανέλθω. Όποτε θεωρείτε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και πάλι ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Και κλείνοντας, για άλλη μια φορά, θέλω να σας πω και το εννοώ ότι σας ευχαριστώ για την βοήθειά σας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Έτσι τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε χάρη στη δική σας υποστήριξη, χωρίς ε, την ε, οποία ε, που θα είχαμε προχωρήσει και αν και το Συμβούλιο και την ίδια στάση με εσά και τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο ρόδινα για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Εγώ, εμεί ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο. Δεν ξέρω δεν ξέρω εάν ισχύουν οι έπαινοι και για μένα. Τέλος πάντων. Ξέρετε υπάρχει και άλλος επιτροπής που περιμένει στην ε, πόρτα να μπει. Τέλος πάντων σας ε, ευχαριστούμε που Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. People should also know that we're seeing you in other fora as well, the clusters and conference of committee chairs and other report backs as well as... Ε, και θα τα πούμε και στα πλαίσια και άλλων συναντήσεων. Ευχαριστούμε και πάλι. Έχουμε και την κυρία Επίτροπο που περιμένει. Uh, Επόμενο θέμα συνάδελφοι. Προχωράμε σε αυτό και είναι εδώ η κυρία Εγώ οπότε παρακαλώ μείνετε στη θέση σα.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 Oh, dear. Dear colleagues, um, we can start point... Ο Πρόεδρος, ας αρχίσουμε με το θέμα υπαριθμών 10. Έκαναμε και ένα μικρό διάλειμμα να με συμπαθάτε. Παρουσίαση του Sir Julian King, Επιτρόπου Αρμόδιου για την Εσωτερική Ασφάλεια από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει εκδώσει διάφορα έγγραφα για το πακέτο κυβερνοασφάλειας, ανθεκτικότητα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις κλπ. Βεβαίως η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται για θέματα εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων ε, στο διαδίκτυο. Είναι καλό που έχουμε κοντά μας τον κύριο Επίτροπο Γνωρίζω ότι πέρασε μόλις από την Επιτροπή Αρμόδια για την, ε, τον αγώνα και βρήκε και χρόνο να έλθει και σε εμά. και εδώ στην Επιτροπή ε, Θεμελιωδών Ελευθεριών. Έχετε κάποια έγγραφα ε, και τις ανακοινώσεις δηλαδή καθώς ε, και άλλα έγγραφα για τα οποία θα μιλήσει ο Επίτροπος. Σου Τζούλιαν, χαίρομαι πολύ που σα βλέπω εδώ και σα παρακαλώ να μου δώσετε το λόγο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλες και όλους εκείνους που είναι κοντά μας σήμερα. Διπλή δόση Επιτροπής λοιπόν Αβραμόπουλος King. Αντιλαμβάνομαι ότι η αφοσίωσή σας στο καθήκον ε, ε, είναι αξιέπαινη. Χαίρομαι που μπορώ να σας μιλήσω για θέματα κυβερνοασφάλειας. Υπάρχουν και παρουσιάσεις οι οποίες ε, διεξάγονται αυτές ε, τις στιγμές γιατί υπάρχει ένας αριθμός επιτροπών που παίζουν σημαντικό ρόλο στην συλλογική αυτή προσπάθεια. Πάντως, ενδιαφέρθηκα πολύ να προσέλθω εδώ ενώπιον ημών στην Επιτροπή Θεμελιδών Ελευθεριών ΛΥΜΠΕ διότι θεωρώ ότι εσείς παίζετε σημαντικό ρόλο επίσης βεβαίως και μαζί με ε, άλλα όργανα και φορείς του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν θεωρώ δε ότι πρόκειται μόνο για τα θέματα που έχουν πιο πολύ άμεση σχέση με το κυβερνοέγκλημα. Νομίζω ότι είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο θεμάτων ασφάλειας που έχουν κεντρική σημασία για το έργο της Επιτροπής σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ε, προσπάθεια, τη δέσμευση και για τον χρόνο σας. Γνωρίζετε, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτός ο διασυνδεδεμένος κόσμος με πολλούς τρόπους συμβαδίζουν και με κάποιους κινδύνους και προκλήσεις που ε, σημαίνει αυτή η διασύνδεση και αν δεν το αναγνωρίσουμε αυτό και αν δεν κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις και να αυξήσουμε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, κινδυνεύουμε να υπονομεύσουμε την αξιοπιστία της διασύνδεσης αυτής, καθώς και την, μοίρα των, ε, την, μάλλον την πίστη των πολιτών μας ε, σε ένα επιγραμμικό μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για την Ευρώπη, αλλά και λόγω των ευρύτερων ε, διακλαδώσεων που έχει το θέμα μας μαζί με άλλους επιτρόπους Έχουμε εργαστεί πάνω σε αυτό ε, το θέμα και έχουμε θέσει επιτάπητο στο θέμα μαζί με τα κρατημέλη και με το Κοινοβούλιο για να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπήρξε μια στρατηγική για το κυβερνο, ε, κυβερνοασφάλεια του 2013 η οδηγία περί της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής που ισχύει είναι πολύ σημαντικό να προστατεύεται η κοινωνία μας, καθώς αναπτύσσονται όλα και περισσότερα επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά τα, η φύση των θεμάτων που συνδέονται με την κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και γι' αυτό και πιστεύουμε πως είναι σωστή η στιγμή να εξετάσουμε και πάλι κάποια από αυτά τα θέματα και να τα συζητήσουμε μαζί σας. Το ίντερνετ των πραγμάτων σημαίνει ε, δεκάδες εκατομμύρια περισσότερες συσκευές θα είναι συνδεδεμένες επιγραμμικά και ε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για να προσπαθήσουν να μας βλάψουν. Ε, οι ε, ε κυβερνοαπειλές καθίστανται πιο στρατηγική σημασίας και ε, αμφισβητούν και τα δημοκρατικά μας, ε, τους δημοκρατικούς μας θεσμούς και μάλιστα εκτός από τον κόσμο της ε, πληροφορικής περνάνε και σε άλλους τομείς, οικονομικούς τομείς. Στα έγγραφα που έχετε νομίζω έχουμε παρουσιάσει την κλίμακα της απειλής από το 2016 4.000 ε, ημερησίες επιθέσεις, 300% αύξηση, πρόσφατες ε, επιθέσεις, ε, WannaCry και άλλοι, δείχνουν πόσο τεράστιο αντίκτυπο μπορεί να έχει μια τέτοια δραστηριότητα. 150 χώρες πλήγησαν ε, άρα λοιπόν σε σχέση με αυτή την κλίμακα της απειλής φτιάξαμε και προτείναμε ένα σύνολο μέτρων ε, που βασίζονται σε τρεις πυλώνες αντοχή, αποτροπή και άμυνα. Και στους τρεις τομείς χρειάζεται να συνεργαστούμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά επίσης και σε ευρύτερο διεθνές επίπεδο. και βεβαίως ε, είναι θέμα του Κοινοβουλίου ε, και του Κοινοβουλίου και ε, ξέρω ότι ασχολείστε και γνωρίζετε τη σημασία της προόδου σε αυτά τα θέματα. Πρώτος από τους πυλώνες είναι η αντοχή. Εμείς χρειάζεται συλλογικά να γίνουμε πιο ε, ανθεκτικοί, δυσκολότερο να μας επιτεθούν και ταχύτερα να μπορούμε να απαντήσουμε όταν ε, γίνονται επιθέσεις. Ως κομμάτι του πακέτου η Κομισιόν προτείνει να δημιουργηθεί ε, μια ισχυρότερη, ένας ισχυρότερος οργανισμός για την κυβερνοασφάλεια με, βάση, την Ενίζα που γνωρίζουμε αλλά με περισσότερες ευθύνες, αρμοδιότητες και πόρους ώστε να έχουμε εξασφαλισμένα συντονισμένη απάντηση όταν υπάρξει επίθεση. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς δουλεύουν όλα αυτά, πώς λειτουργούν όλα αυτά και να επεκτείνουμε αυτού του είδους την προστασία πέρα από τους κρίσιμους τομείς της υφιστάμενης νομοθεσίας αλλά και σε άλλους τομείς κινδύνου όπως οι δημόσιες ε, σχέσεις, το, καλά, δημόσιες υπηρεσίες και, και νοσοκομεία. Θέλουμε να υπάρχουν εβδομάδες γρήγορης ανταπόκρισης με τους κατάλληλους πόρους και στελέχωση. Πρέπει επίσης να παίξουμε ρόλο στην εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής διάστασης, ενός ευρωπαϊκού πλαισίου μάλλον πιστοποίησης που θα εξασφαλίζει πως η ασφάλεια είναι σωματωμένη στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, δηλαδή ασφάλεια μέσα στο σχεδιασμό. Ε, ο οργανισμός αυτό εξασφαλίσει επίσης ότι δεκάδες δισεκατομμύρια νέα συνδεμένα προϊόντα θα έχουν αντοχή ε, στις επιθέσεις πριν να τοποθετηθούν στην αγορά και μετά. Γιατί η απειλή ε, εξελίσσεται. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ε, ε, ευρωπαϊκών διαστάσεων σχέδια επιστοποίησης επί τη βάση των όσων ήδη έχουμε. Ήδη υπάρχουν κάποια καλά σχέδια, αλλά να δημιουργηθεί και ένα σύνολο πανευρωπαϊκών κανόνων, απαιτήσεων και στάνταρ, ώστε οι πολίτες μας να γνωρίζουν και την ε, τα, τις υπηρεσίες που μπορούν να, να εμπιστευθούν και να μπορούν να γνωρίζουν, ε, να, να έχουν μάλλον μια σταθερή ποιότητα. Λοιπόν, οι νόμοι και οι, ε, οι κανονισμοί είναι σημαντικοί, αλλά και το ίδιο είναι σημαντική είναι και η κουλτούρα, γιατί Πολλές φορές ε, οφείλεται ε, η επιθέσεις στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Ξεκινά η κυβερνοασφάλεια στο σπίτι με την κυβερνογενή ασφαλή σκοδική ε, ασφαλές περιβάλλον. Πρέπει σοβαρά να το λάβουμε υπόψη ως άτομα και να βοηθήσουμε τον κόσμο να αναλάβει αυτές τις ευθύνες και οι επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας πρέπει να υιοθετήσουν ένα κατάλληλο χώρο, να έχουν κατάλληλα προγράμματα ασφάλειας, να τα ανανεώνουν τακτικά ώστε να ανταποκρίνονται στο εξελισσόμενο ε, τοπίο της ε, κυβερνοεγκληματικότητας. Τώρα η αντοχή σημαίνει και η δημιουργία δεξιοτήτων, η απόκτηση δεξιοτήτων. Έχουμε 350.000 κόσμο που λείπει, που θα λείπει μάλλον μέχρι το 2022. Οι ανάγκες είναι μεγάλες, πρέπει που κατά προτεραιότητα να συμπεριλαμβάνονται αυτού του είδους οι σπουδές στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι γεγονός ότι πολλοί κατασκευαστές, ευρωπαίοι κατασκευαστές εξαρτώνται από την αγορά κρίσιμης τεχνολογίας εκτός Ένωσης. Οπότε θέλουμε να οθήσουμε τις ευρωπαϊκές ε, βιομηχανικές δυνατότητες, παραγωγικές δυνατότητες και τα πρώτα βήματα έγιναν με την εταιρική σχέση ιδιωτικού με ε, δημόσιο τομέα, ΣΔΙΤ, για την κυβερνοασφάλεια που θα κινητοποιήσει πολλά εκατομμύρια μέχρι το 2020, αλλά στην Αμερική δαπανώνται 17 δις δολάρια μόνο φέτος για αυτό το θέμα. Θέλουμε να προχωρήσουμε λοιπόν περισσότερο, προτείνουμε πανευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας για να ενισχυθούν οι δυνατότητες ολόκληρη την Ευρώπη και παράλληλα μια νέα ευρωπαϊκή έρευνα ένα κέντρο μάλλον, πανευρωπαϊκό κέντρο έρευνας και δεξιοτήτων στην κυβερνοασφάλεια, ώστε να αποτελέσει ένα κόμβο για να βοηθήσει και να στηρίξει τις ευρωπαϊκές εταιρείε. Θα το υποβάλουμε αυτό από το χρόνο. θα φτιάξουμε μια πιλωτική φάση που θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Ενίσχυση της αντοχής σημαίνει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε όταν συμβεί το χειρότερο. Όπως οι πρόσφατες επιθέσεις έδειξαν, κάποια συστήματα έχουμε φτιάξει, αλλά πρέπει να γραφτούν περισσότερα. Πρέπει να φτιάξουμε λοιπόν ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα για το πώς ανταποκρινόμαστε σε σοβαρέ κρίσει που πρέπει να το ελέγξουμε και να το επικυρώσουμε με τα κράτη-μέλη και τους, όλους τους Το να είναι πιο δύσκολο να μα επιτεθεί κανεί, είναι σημαντικό τμήμα τη απάντησης, αλλά δεν είναι ολόκληρη η απάντηση. Χρειάζεται και αξιόπιστα ε, μέτρα αποτροπής για τους δυνητικούς ε, δράστες, είτε είναι εγκληματίες, είτε είναι, είναι ε, κρατικοί εχθρικοί δράστες, είτε μη κρατικοί δράστες ε, εχθροί. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να εστιάσουμε στην αύξηση των πιθανότητων να συλληφθούν με αξιόπιστες και, αποτρο... απο... ε, και ποινές αποτροπής. Εντοπισμός, ανεχνευσιμότητα, δικαστική έρευνα και ποινική δίωξη. Πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και με τον ιδιωτικό τομέα σε όλα αυτά τα θέματα. Οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει επίσης να συμβαδίζουν με την τεχνολογία και επίσης να μοιραστούν εμπειρογνωμοσύνη στις ε, ε κυβερνοέρευνες και πάλι προτείνουμε την Europol ως πιθανό κόμβο για την αντιμετώπιση επιθέσεων. Υπάρχουν προκλήσεις στην πρόσβαση των ψηφιακών αποδείξεων, όπως ξέρετε, που το έχουμε ξαναπεί, αλλά είναι ιδιαίτερα ε, σημαντικό εδώ. Θέλουμε λοιπόν να δράσουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε κάποιους από τους φραγμούς ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτό του είδους τις αποδείξεις της ε, διώξης μας. Ε, οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι διασυνοριακές εξορισμού και η εργασία των εισαγγελέων και των ε, ανακριτών είναι πιο περίπλοκη γιατί αυτή πρέπει ακόμα, να, ακόμα περιορίζονται από τα εθνικά σύνορα οπότε μαζί με την Επιτροπό Γιούροβα θα υποβάλουμε ένα σύνολο προτάσεων στις αρχές του χρόνου, ώστε να έχουμε μία μοναδική πρόσβαση για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και για τα κυβερνοεγκλήματα και κυβερνοεπιθέσεις. Ε, τονώνουμε τη δυνατότητά μας για διώξεις και για επιβολές κυρώσεων για ορισμένες μορφές κυβερνοεγκλήματος, όπως ας πούμε για την παιδική ε, ε, σεξουαλική παρενόχληση προτείνουμε την αντιμετώπιση των απατών πληρωμής που είναι όλο και περισσότερο ψηφιακό ε, αδίκημα απάτες για όλες τις όλα τα εμβάσματα, όλες τις πληρωμές, ακόμα και για εικονικά νομίσματα συγκεκριμένες ποινές και να διευκρινίσουμε το πεδίο της δικαιοδοσίας των κρατών μελών ώστε τα διασυνοριακά εγκλήματα για δικήματα να μπορούν να διωκόνται πιο εύκολα. Επίση, πολιτικέ απαντήσεις, ας πούμε, μέσα από τις αμυντικέ δυνατότητες των κρατών μελών, πρόκειται για γιατί εδώ έχουμε ένα, σαφώς ένα στοιχείο άμυνας και θέλουμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να διευνήσουμε το πεδίο της χρήσης κονδυλίων από την άμυνα της Ένωσης για να ενισχύσουμε τις δυνατότητες κυβερνοάμυνας. Τέλος πρέπει να οθήσουμε τις διεθνείς διαδικασίες για να συμφωνήσουμε για πρότυπα ε, κρατικής συμπεριφοράς για τη δημιουργία ε, μέτρων ε, οικοδόμησης εμπιστοσύνη στο κυβερνοχώρο. Ε, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τον Ιούνιο συμφώνησε για ένα, μια εναργαλειοθήκη κυβερνοαντιμετώπισης, κυβερνοαπάντησης σε απειλές όπου περιλαμβάνονται και κυρώσεις. Πρέπει να δουλέψουμε λοιπόν με βασικούς διεθνούς, διεθνείς εταίρους για αυτά τα θέματα. Πρέπει να συνεχίσει λοιπόν και η εργασία και στον ΟΗΕ, η συνεργασία μάλλον με τον ΟΗΕ, να φτιάξουμε όσο γίνεται περισσότερη υποστήριξη ε, και αντοχή στις γειτονικέ και άλλες τρίτες χώρες, να αυξηθούν τα επίπεδα κυβερνοασφάλειας παγκοσμίω. Αλλά επίσης πρέπει να ενεργήσουμε ώστε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με τον ΝΑΤΟ είναι ένας τομέας όπου η κοινή δήλωση που υπογράφει το, στη Βαρσοβία πέρυσι μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ ε, παραθέτει διάφορες φιλοδοξίες. Τώρα πρέπει να δοθεί συνέχεια. Έχει γίνει πρόοδος ε, για πρώτη φορά τα επιτελεία ΝΑΤΟ και Ένωσης οργανώνουν και κρεών ασκήσεις από κοινού. Αυτό το στηρίζω και ε, θα ήθελα μαζί σας να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε ώστε να εμπλουτίσουμε τις προσεγγίσεις μας στην αντοχή και στην αναχέτηση κυβερνητικών, ε, κυβερνοαπειλών και κυβερνοεπιθέσεων. Επίσης, υιοθετήσαμε ένα κοινοθένα για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου online, γιατί αυτό, και αυτό το αναφέρω γιατί συνδέεται με αυτά τα θέματα. Εκείνα τα ανακοινωθέν παρουσιάζει κατευθύνες γραμμές για τη στήριξη των πλατφορμών online ε, να δημιουργήσουν ε, δραστήριες δραστήριο εντοπισμό παρανόμου περιεχομένου, δηλαδή ε, ε, λόγω μίσους, ε, διακρίσεων και ε, τρομοκρατικές, μάλλον, παρακήρυξη τρομοκρατικές ενέργειες. Εδώ δεν λέμε τι είναι παράνομο ή τι είναι παράνομο, αλλά αυτό παρουσιάζεται αλλού, χωριστά σε άλλη νομοθεσία. Αλλά υπάρχει υλικό online ακόμα και σε γνωστές πλατφόρμες που ε, την τρομοκρατία ή δείχνουν στον κόσμο πώς να κάνει τρομοκρατικές απόπειρες. Πρέπει λοιπόν οι εταιρείε να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να απαγορεύσουν τέτοιο είδους υλικό. Αυτό το ανακοινωθένει το πρώτο Τώρα το τι θα κάνουμε μετά εξαρτηθεί από το πώς θα ανταποκριθούν αυτές οι, πλατφόρμες. Θα παρακολουθήσουμε την πρόοδο για το υπόλοιπο του έτους και στις αρχές του επόμενου χρόνου θα αξιολογήσουμε αν έχει γίνει πρόοδος και αν, να αποφασίσουμε αν χρειάζεται περαιτέρω δράση η νομοθεσία. Το πρώτο στοιχείο αυτού του φιλόδοξου πακέτου είναι μαζί τώρα, μαζί με μια ευρεία ομάδα συνεπιτρόπων που εργάζονται για αυτά τα θέματα, σε αυτή την Επιτροπή αλλά και σε άλλες αρμόδιες επιτροπές να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όπως ανακοινώσαμε, ετοιμάζονται περαιτέρω προτάσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ηλεκτρονικές μαρτυρίες, και όλα μαζί νομίζω συμβάλλουν σε, μια, σε ένα στρατηγικό στόχο που είναι να ενισχυθεί η κυβερνοαντοχή μας ε, για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και... ακούσουμε τους κύριε Μετσόλα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και συμπαθέτε με ε, διότι πρέπει να φύγω αμέσως μόλις ε, ε, σας μιλήσω γιατί πρέπει να βρίσκομαι σε μια άλλη επιτροπή. Μπορούμε και στις δύο. πάντως ευχαριστούμε που ξανά ήρθατε να μας δείτε. Ευχαριστούμε για όλα όσα κάνατε αυτή σας την πρωτοβουλία για να βελτιώσετε την κυβερνοασφάλεια και το κυβερνοέγκλημα μας ε, οδηγεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Είναι η 21 ου αιώνα η πιο σημαντική μας πρόκληση, γιατί όλοι έχουν ε, φύγει χωρίς καμία εξαίρεση από αυτό. Και ε, οι υποδομές μας μπαίνουν σε δοκιμασία. Έχουμε κάποιου κινδύνου οι οποίοι γίνονται όλο και πιο έντονοι, άρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα σύστημα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε διοικητικέ αρχέ να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από του ε, εγκληματίε που θέλουν να εκβιάσουν, θέλουν να επιτεθούν. Οπότε εμεί ε, θεωρούμε πάρα πολύ θετική αυτή τη δέσμη μέτρων. Θέλουμε πάντω να θεωρήσουμε να, ότι είναι πολύ θετικό αυτό που προβλέπετε για την ΕΝΗΣΑ, για αυτή την μόνιμη εντολή, ούτω ώστε τα κρατημέλια να μπορούν να κάνουν μια πρόληψη, να μπορούν να αντιδράσουν στι κυβερνοεπιθέσει. Θα πρέπει να έχουμε συμβατότητα οι υπηρεσίε του κάθε ε, κράτου με τα άλλα, θα πρέπει να έχουν καλή προοικοδότηση αυτέ οι υπηρεσίε, ούτω ώστε να αναπτύξουν τι δυνατότητε για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον ολοένα μεγαλύτερο φόρτο εργασία και να κάνουν τη δουλειά του για το κυβερνοέγκλημα. Ε, επίσης είναι θετική η πρόταση για μια οδηγία καταπολέμησης της ε, απάτης. Τώρα θα καλυφθούν περισσότερα εγκλήματα ε, εις βάρος του συναλλαγών, εις βάρος της πληροφορικής και με τα ηλεκτρονικά τα κατηδέαν τέλο πάντων νομίσματα. Ε, είναι ένα μεγάλο βήμα αυτό προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτό θέλαμε από σα τέτοιε πρωτοβουλίε. Επίση, αυτού του είδου το πλαίσιο θα μας επιτρέψει να αντιδρούμε καλύτερα, πιο γρήγορα και σε μεγάλες κλίμακες κυβερνοεπιθέσεις. Ε, αυτά τα θέματα πρέπει να καλύψουμε και έτσι να υπάρχουν έρευνες, δίωξη, κυρώσεις για τις, αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις, το κυβερνοέγκλημα. Χρειάζεται άρα συνεργασία για την καταπολέμηση του κλίματος και έτσι θα προστατεύσουμε τον κόσμο περισσότερο και κυρίως τους ανηλίκους, αλλά τις επιχειρήσεις τα δίκτυά τους και την υποδομή τους. Οπότε θα πρέπει να μπορέσουμε αποτελεσματικά να απαγορεύσουμε το παράνομο περιεχόμενο από κάποιους ε, παρόχους υπηρεσιών και ευνηδιαστικά. Μέχρι τις 4.30 έχουμε συνάδελφοι, παρακαλώ, ένα δίλεπτο μόνο. Ευχαριστούμε Επίτροπε, εκεί που ήρθατε στο Κοινοβούλιο, που μας μιλήσετε για αυτά τα σημαντικά πολύ σημαντικά ακούσαμε. Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο πολύ μικρά ε, παραδειγματάκια. Ότι δηλαδή πολλοί συμπολίτε μας δεν έχουν ιδέα για το τι γίνεται στον ψηφιακό κόσμο. Α, βλέπουν μια εφαρμογή, λένε ας την κατεβάσω, αλλά δεν ξέρουν τι γίνεται δεν ξέρουν ότι παρακολουθούνται. Δεν τους νοιάζει από ποιον παρακολουθούνται και για ποιο λόγο. Δεν σκέφτονται ότι ίσως κατεβάζοντας την λόγο εφαρμογή θα κατεβάζουν μαζί και κάποιο ιό. Μια μέρα όμως λένε «Α, για να δούμε, για να βρω κάποιες πληροφορίες ε, τις πάρω στη δουλειά, να δουλέψω εκεί, παίρνουν τα δεδομένα σε ένα USB, τα πάνε στη δουλειά τους και εκεί υπάρχουν κάποιες σοβαρές υποδομές, οπότε ο ιός μολύνει και το χώρο δουλειάς. Αυτό θα πρέπει να μας νοιάζει. Μιλώντας για κυβερνοασφάλεια, θα πρέπει και στις χώρες μας να ενημερώνουμε γιατί εδώ και χρόνια δεν το έχουμε καταφέρει. Τα μίντια θα πρέπει να το προσέξουν. Άλλο ένα παραδειγματάκι να σας αναφέρω. Όταν μιλούμε για ασφάλεια των ε, δεδομένων έχουμε την τεχνολογία RFID. Μια μέρα ήμουν σε ένα σούπερ μάρκετ, δεν είχα μαζί μου αρκετά μετρητά και πήρα την ε, κάρτα μου πήγα να τη βάλω στη συσκευή, στη σχισμή και μου είπαν όχι δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται απλώς πλησιάστε την κάρτα σας στη συσκευή και θα πληρώσετε ναι ωραίο αυτό απλό όμως έτσι οι εγκληματίες μπορούν αν είναι κοντά μου, πίσω μου ας πούμε στην ουρά να διαβάσουν τα δεδομένα μου Άρα χρειάζεται αυτό το gadget το οποίο μπλοκάρει και άρα για όλα τα προβλήματα που έχουμε θα πρέπει αντιστοίχω να σκεφτόμαστε τις λεπτομέρειες, να μην τα ξεχνάμε. Γιατί στο παρελθόν μάθαμε ότι όταν μιλούμε για οργανωμένο έγκλημα δεν είναι πια δουλεμπόριο, λαθροδιακίνηση προσώπων, ναρκωτικά κλπ αλλά πολλέ φορέ αυτά που νομίζαμε ότι είναι μικρά δικήματα, αυτά γίνονται μεγάλα γιατί γίνονται σε μεγάλη κλίμακα από τι συμμορίε. Για αυτή την τεχνική που είπατε, για αυτό το, το γκατζετάκι που προστατεύει, καλά εγώ δεν είμαι τόσο περιβολικός όπω εσεί αλλά το ξέρω, το ξέρω. Έχετε δίκιο. Δεν ξέρω, το έχει ο Επίτροπος για την ε, κυβερνοασφάλεια, αυτό το ρίθιτο ποτέ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να το τύχει. Καλό είναι για προστασία. Σαργεντίνη, please. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Κίνγκ και οι υποφαινομένοι συνευρισκόμεθα στον ίδιο χώρο, αλλά έχω να σας αναφέρω τα εξής, ε, αν δεν έχετε αντίρρηση. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι θέλετε να αντιμετωπίσετε το, τα προβλήματα που έχουν τα κάτι ε, νομίσματα. Έχουμε και την οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος, οπότε είπαμε ότι θα πρέπει να δοθεί ένας ορισμός του τι είναι αυτά τα, τα, τα ψηφιακά νομίσματα, τα virtual νομίσματα. Άρα θα πρέπει να το το θέμα στην οδηγία ε, αυτή μου, αν μας αναφέρεται θα βοηθήσει πάρα πολύ. Άλλο τώρα. Τι γίνεται με αυτές τις κερκόπορτες, ας πούμε, backdoors και zero days, γιατί στις ε, ποινικέ έρευνες υπάρχει πρόβλημα. Θα θέλαμε να μπορούν οι διοικητικέ αρχές να κάνουν τη δουλειά του, αλλά δεν θέλουμε από την πίσω πόρτα να μπορούν να ερευνήσουν τα δεδομένα που υπάρχουν. Αυτή την zero day. Το θέμα είναι να γίνονται όλα αυτά σύνομα. Να είναι νόμιμη δηλαδή οι συνθήκε της έρευνας. στις κάτω χώρες μας απασχολεί το θέμα αυτό. Τώρα όσον αφορά το να αφαιρείται από σελίδες του ίντερνετ περιεχόμενο που αφορά εγκλήματα και τρομοκρατία. Και αυτό θα πρέπει να οριστεί, να περιχαραγωθεί. Υπάρχουν και διαφορές στη ρύθμιση από χώρα σε χώρα. Πολλές φορές αυτά τα αναθέτουμε σε κάποιους παρόχους υπηρεσιών ίντερνετ. Όμως αυτό είναι δουλειά για τις κρατικές αρχές. Δεν θα έπρεπε να έχουμε υπεργολαβίες για αυτή τη δουλειά. Θα πρέπει να εναρμονιστούν επομένω και οι ορισμοί και τα σχετικά μέτρα και να μην αναθέτουμε σε εμπορικές εταιρείες αυτά τα καθήκοντα αυτές τις δουλειές. Ζεράρ Ντεπρέ. Ah, merci, euh, Euh, l'indulgence de... Κύριος στις δικές γνώσεις, γιατί εγώ δεν τα ξέρω τα θέματα της ασφαλείας. Και συγγνώμη κύριε Επίτροπε, γιατί μπήκα στην αίθουσα την ώρα που μας μιλούσατε. Όχι, εγώ δεν είμαι το ίδιο παρανεκός και υπερβολικός όπως ε, ο πρόεδρος αλλά σας είπα δεν τα ξέρω πολύ καλά και προβληματίζομαι και έχω να σας πω επίτροπε μία σκέψη μου να κάποιος που δεν τα ξέρει τα θέματα όπως εγώ μπορεί να πει ότι να, το ίντερνετ ο χώρος του ίντερνετ είναι χώρος χωρίς σύνορα και όταν έχουμε επιθέσεις δεν έχουν σύνορα γιατί μπορεί οι στόχοι να είναι ταυτόχρονα πολλοί σε διαφορετικά μέρη, σε ιδιωτικό χώρο, σε δημόσιο χώρο κλπ. Αυτό θέλω να μου ξεκαθαρίσετε. Στις προτάσεις της Κομισιόν προβλέπονται κάποιες δυνατότητες, δημιουργία δυνατοτήτων κυβερνό αμήνης. Για παράδειγμα, μάθαμε ότι στην ε, Γαλλία ότι συγκροτήθηκε κάποια υπηρεσία για την προστασία, για την άμυνα σε επίπεδο κυβερνοσφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια που δεν είναι τόσο ξεκάθαρα περιχαρακωμένα τα πράγματα και τα σύνορα αυτή του προβλήματος γίνεται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να έχουμε μια υπηρεσία αυτόνομη. Μίλησατε για 350.000. Είναι πάρα πολλοί αυτοί. Αυτούς να τους βάλουμε σε κάποια υπηρεσία κεντρική, πανευρωπαϊκή αυτή να είναι top η υπηρεσία υπερ αποτελεσματική. Ε, αυτό θα ήταν οικονομία να μην έχει και το κάθε κράτος τους δικούς του. Μου λένε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Προστασία των Δικτύων ε, δούλευε εντατικά. Όμως, αν δεν κάνω λάθος, κάνουν διαγωνισμό κάθε χρόνο αυτή. Ε, διαγωνισμό για να διαγωνιστούν οι, οι ειδικοί στα θέματα κυβερνών ασφαλείων. Κάτι άλλο που με απασχολεί. Καταπολέμηση τρομοκρατίας, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Οι κυβερνο Δηλαδή συγκεκριμένα εννοώ κάποιους Διαστραμμένους που έχουν στόχους τους ανηλίκους και μέσω του ίντερνετ κρύβονται κλπ. λοιπά Τι μπορούμε να κάνουμε από πλευράς νομοθετικής. Ε, υπάρχει θέμα από τις δικές μας χώρες αλλά μέχρι και τον Καναδά. Ο επόμενος. Ευχαριστώ. Επίτροπε. Εδώ το μας είπατε. Ευχαριστούμε για όλα σε αυτές τις προτάσεις, αυτό το πακέτο κυβερνοασφάλειας. Ε, βέβαια και όλο και αυξάνεται ο κίνδυνος. Από το 16 είχαμε πάνω από 4.000 επιθέσεις του λεγόμενου ransomware και από το 2015 αυτό ήταν αύξηση κατά 300% και 80% των εταιριών στην Ευρώπη εφήγησαν από αυτές τις επιθέσεις. Έχω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα σε σχέση με όσα μας είπατε για το δέσμο μέτρο. Συντονισμός και συνεργασία. Είναι σαφές. Πρέπει να έχουμε στην Ενίσα νέα εντολή να έχουμε καλύτερη, αναβαθμισμένη συνεργασία τον μελών. Επίσης, περισσότερη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, Europol, ENISA, EASA κλπ. Είναι πολλές πληροφορίες, είναι πολλά τα δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρχει η σωστή και ταχεία ανάλυση Επίσης, πιο κάτω μας είπατε ότι άρχισε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Πολύ σημαντικό. Γιατί δεν μιλούμε μόνο για μη στρατιωτικές απειλές. Έχουμε και το θέμα της άμυνας και του υβριδικού πολέμου. Ελπίζω όμως ότι κάνουμε μία αρχή και ότι θα έχουμε Υπάγειο συνεχή χαρακτήρα αυτή η συνεργασία. Πολύ σημαντικό αυτό. Συμφωνώ 100% με την Μπίρκετ. Θα πρέπει πρώτα-πρώτα το πρόβλημα να το επισημάνουν, το συνειδητοποιήσουν όλοι. Θα πρέπει κάποια θέματα να τα αντιμετωπίσουμε και ως άτομα, αλλά να υπάρξει ευρία διάδοση του φαινομένου πιστοποίηση τώρα και την κατοθεσία. είναι σαφέ σε όλα τα έγγραφα τη Κομισιόν το που πρέπει να, προς τα που πρέπει να αλλά να μην έχουμε ενιαία λύση για όλους. Πρέπει να συνεργαστούμε με πολλούς τομείς. Άρα, ναι, δικαιοθεσία αλλά θα πρέπει να κινηθούμε όπως ταιριάζει στον κάθε συνομιλητή μας. Και έτσι να προκύψουν λύσεις ξεκάθαρες. Τώρα, όσο να βρω τι θα κάνουμε για κάποιες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνο, Πρώτα πρώτα να δούμε το πώς οι οδηγίες πρέπει να δώσουν, πώς θα αποδώσουν και μετά να αναζητηθεί η λύση, ίσως ε, νομοθετικά. Αλλά τι λέτε γι' αυτό. Σε πολλές χώρες έχουμε διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή, οι οδηγίες, οι κατευθυντήριες γραμμές που δίνουμε θα εφαρμοστούν και θα, θα γίνουν αποδεκτές με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να εμπλέξουμε όλους. Ευχαριστώ. Thank you very much, Commissioner. Ευχαριστώ εσείς Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ενημέρωση για, το, για τις σημαντικές αυτές νέες εξελίξεις. Και... Βλέποντας το έργο σας βλέπω πολλά καλά στοιχεία όχι μόνο για την κυβερνοασφάλεια, αλλά είναι και σημαντική και η εκπαίδευση του κόσμου. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Υπάρχει μια διασύνδεση εδώ, όπως έλεγε προηγουμένως ο βουλευτής κ. Μπόνι. Διότι προκαλείται σύγχυση από την έλλειψη ορισμού τι ακριβώς είναι το κυβερνό έγκλημα, τι σημαίνει κυβερνό ασφάλεια και αυτά που είπατε στην ομιλία σας ε, κάπως ε, τυχαία ψηφιακή ασφάλεια και ψηφιακό έγκλημα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία έχουν σχέση με την ψηφιακή ασφάλεια των προσώπων. Και βεβαίω αυτά δεν μπορούν να λυθούν μόνο με ρύθμιση. Χρειάζεται νέα ποινική νομοθεσία. Διότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία εμφανίζονται στο γενικότερο περιβάλλον και έχουν σημαντικότατες σοβαρές επιπτώσεις στους ανθρώπους, στην υγεία τους, στην ασφάλειά τους, στην ασφάλεια του σπιτικού τους και ούτω καθεξής. τι συνεργασία έχετε με την, με την Επίτροπο Γιώροβα, διότι χρειαζόμαστε νέες ποινικέ διατάξεις στους ποινικού κώδικες. Πρέπει να προσθεθούν νέα κεφάλαια που θα αναφέρονται στο έγκλημα στον ψηφιακό χώρο. Όχι δηλαδή μόνο το κυβέρνο έγκλημα με τη στενή έννοια. Κάτι που είναι επίγον και που σας ζητούμε εμείς αλλά και από την Επίτροπο κυρία Γιώροβα να το βάλετε στο θεματολόγιο είναι το πρόβλημα των παιδιών. Το αναφέρθηκε και πριν. Χρειάζεται να μπει στην νομοθεσία κάτι για την ανάγκη ειδική προστασία των παιδιών. Αντιμετωπίζουμε όμως νομικές δυσχέρειες στην προσπάθεια αυτή. Δεν βρήκαμε δηλαδή το κατάλληλο νομικό έδαφος για να τα βάλουμε τα πράγματα αυτά. Για παράδειγμα, για τα παίγνια. Για τα παίγνια. Εννοείται ηλεκτρονικά παιχνίδια πρέπει με κάποιο τρόπο να προληφθούν οι κίνδυνοι για τα παιδιά. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία οδηγούν σιγά σιγά τα παιδιά στην αυτοκτονία. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ποινικοποιηθούν. Είναι πολύ εξειδικευμένοι χώροι αυτοί. Ε, σας ζητώ όμως να εγκύψετε σε αυτά, διότι χρειάζεται η υψηλή προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, όχι μόνο στην χρήση των τεχνολογιών, αλλά και σε τέτοιου είδους καθημερινές δραστηριότητες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το άλλο που βλέπω κάπως να λείπει στο καλό έγγραφο που υποβάλατε είναι αυτή η διασύνδεση μεταξύ e-privacy και security. Αντιμετωπίζονται πιέσεις, αντιμετωπίζονται προκλήσεις για τη δημιουργία μια τεχνητή σύγκρουση κατά κάποιο τρόπο μεταξύ προστασίας προσωπικής σφαίρα και τη ασφάλειας. Είναι πολύ διασυνδεδεμένα αυτά τα πράγματα, προσωπική σφαίρα και ασφάλεια. Εγώ θα ήμουν πολύ ικανοποιημένη να δω να αναπτύσσονται τέτοια θέματα μια πιο θετική διασύνδεση και μια συνεργασία ανάμεσα στους χώρους αυτούς που καλύπτουν και τα δύο θέματα, δηλαδή και την προσωπική σφαίρα και την προστασία της προσωπικής σφαίρας και την ασφάλεια. Δεν μιλώ τόσο για security όσο για safety, δεν μιλώ τόσο δηλαδή για ασφάλεια απέναντι σε κάποιο ατύχημα, αλλά σε προστασία. Ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπατε. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθο, λέει ο πρόεδρο Κλοντ Μωράε. Έχω ακόμα την τελευταία παρεμβαίνουσα που είναι η κυρία Σπινέλη. Α, και η κυρία Γκόμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Επίτροπε, έχω κάποιες ερωτήσει για θέματα που με ενδιαφέρουν, κυρίως ως εισηγήτρια για την ε, ελευθερία, ελευθεροτυπία και με ενδιαφέρουν αυτά τα μέτρα λόγω των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν ε, περί αυτών, αυτού του είδους την ελευθερία. Το πρώτο ερώτημα που ήθελα να θέσω είναι ότι δεν θα ήθελα αυτή η κίνδυνοι για τους οποίους εσείς μιλήσατε για την κυβερνοασφάλεια, δεν θα ήθελα να παρουσιάζονται δυσανάλογα μεγάλοι. Το λέω γιατί αναφέρατε το μοντέλο των ΙΠΑ 17 δις δολάρια φέτος ε, ως πρότυπο, ως παράδειγμα προς μίμηση. Εγώ έχω αμφιβολίες για το αμερικανικό πρότυπο για αυτά τα θέματα. Αν σκεφτούμε στην μανία που έχουν για την ασφάλεια από τις τελευταίες εκλογές, για κυβερνοεπιθέσεις που, για τις οποίες δεν υπάρχει για την ώρα καμία απόδειξη. Οπότε ανοχή και αποτροπή ναι, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό να ορίσουμε ξεκάθαρα ποιο είναι το παράνομο περιεχόμενο που περνά μέσα από το ίντερνετ και διαβάζεται μέσα από το ίντερνετ ακριβώς επειδή η ελευθερία έκφρασης ε, δεν θα πρέπει να παραβιάζεται. Και πρώτα απ' όλα λοιπόν όταν μιλάμε για, για ποινικέ προθέσεις εγκληματικέ προθέσεις, οι εχθρικές ε, προτάσεις, ε, δεν νομίζω πως είναι το ίδιο. Η εχθρικότητα δεν είναι απαραίτητα και εγκληματικότητα. Ίσως να μην ε, κατάλαβα καλά. Πάντως, Πρέπει να είναι σαφές ότι ποια είναι τα παράνομα περιεχόμενα και να κλείσουμε όσον αφορά την ανάγκη συνεργασία των πλατφορμών ίντερνετ για την απομάκρυνση του παράνομου περιεχομένου. Και αυτή η συνεργασία μπορεί να είναι και επικίνδυνη για την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία τύπου. Εάν σκεφτεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο η Google αποφάσισε να ε, αφαιρέσει από το σύστημα επιλογής ε, στην αναζήτηση site και πληροφοριών, να απομακρύνει λοιπόν τις πληροφορίες για site τα οποία θεωρεί ακραία και όχι εγκληματικά. Και εδώ πάλι δεν είναι το ίδιο. Ακραίος δεν θα πει, εξτρεμιστής δεν θα πει ε, ε εγκληματίας. Είναι απόφαση λοιπόν της Google, αλλά όπως είπα, τη θεωρώ πως είναι επικίνδυνη με ε, η συνεργασία με τους παρόχους του ίντερνετ για την ελευθερία. Η κυρία Άννα Γκόμες, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ερωτώ. Μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσει και να ζητήσει από τις χώρες μέλη, για παράδειγμα, να κάνουν μια προσπάθεια να εντοπίσουν τα ευάλωτα σημεία των ε, συστημάτων τους. Δηλαδή, πόσες εταιρείες ελέγχονται από κινέζικες εταιρείες, όπως η Huawei, Huawei, οι οποίες απαιτούν τα δεδομένα να αποθηκεύονται στην Κίνα, για δικούς τους λόγους. Μπορεί να μιλήσει κανείς πράγματι για κυβερνοασφάλεια όταν δεν υπάρχει έννοια, δεν υπάρχει καμιά ιδέα για τα τροτά σημεία των συστημάτων μας. Ένα παράδειγμα ήταν αυτό. Sorry, colleagues, I'm having discussions about... Εξακολουθώ να ασχολούμαι με τις υποθέσεις της επόμενης εβδομάδας, να με συμπαθάτε, λέει ο πρόεδρος Μωράες. Θα παρακαλέσω τώρα τον Επίτροπο να καταβάλει προσπάθεια να κάνει το αδύνατον, δηλαδή να απαντήσει Έρχεται όμως και άλλη ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την παρακαλώ να έχει κάποια υπομονή ώστε να μπορέσει ο Επίτροπος Αρμόδιος για την Ασφάλεια να απαντήσει. Σε Τζούλιαν, σε παρακαλώ προσπάθησε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την δέσμευσή σας για τα θέματα αυτά και την υποστήριξη. Και δείχνουν οι ερωτήσεις σας ότι η Επιτροπή σας ε, παρακολουθεί πολύ προσεκτικά το follow-up στις ανακοινώσεις. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να απαντήσω πραγματικά σε όλες τις ερωτήσεις. Αν δεν μπορέσω, επανέλθετε. Για την ερώτηση που νομίζω έθεσε η κυρία Μεζόλα και την οποία επανέλαβε ο κύριος Μπόνι. Είμαστε δηλαδή βέβαιοι ότι με τις διάφορες προτάσεις κάνουμε κάτι το σκόπιμο, το οποίο έχει και μια συνοχή με τις ε, προτάσεις ε, που κάνουν όλοι οι φορείς. Ελπίζω, ελπίζω. Αυτό ε, προτιμώ να σκέπτομαι ότι αυτό κάνουμε. Βέβαια, είναι περίπλοκο αυτό που κάνουμε. Αυτό που λέμε βασικά όμως είναι ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε τον οργανισμό ΕΝΙΣΑ που κάνει το reporting, κάνει την σύνταξη εκθέσεων, τις πιστοποίησεις και αντιμετωπίζει τα προβλήματα ασφάλειας. Χρειάζεται να ενισχυθεί λοιπόν σημαντικά ο ΕΝΙΣΑ. Όμως υπάρχει και ένα θεματολόγιο σχετικά με την ασφάλεια του μέλλοντος και εκεί χρειάζεται να πατήσουμε τον γκάζι πραγματικά για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο με ένα βασικό άξονα έρευνας γύρω από τον οποίο θα περιστρέφεται το δίκτυο αυτό υπάρχει μια σημαντική πρόκληση κυβερνοεγκλήματος. Άρα το να βασιστούμε στον ρόλο της Ευρωπόλ, η c που αναγνωρίζεται και διεθνώς ως κέντρο υπεροχής για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος, αυτό που θέλουμε είναι να ενισχύσουμε το έργο αυτό και υπάρχει και ένα στοιχείο άμυνας και από αυτού του στοιχείου άμυνας αυτό που λέμε είναι ότι σε πρώτο βαθμό σε πρώτο βαθμό, η κυβερνοάμυνα υπό την αυτή έννοια είναι κάτι το οποίο κάνει χωρίς μέλη. Θέλουμε όμως να διερευνήσουμε τις δυνατότητες στήριξης των χωρών μελών. Μαζί δηλαδή με τις χώρες θέλουμε να αναζητήσουμε δυνατότητες χρήσης του καινούργιου ε, ε, Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου για να χρηματοδοτήσουμε και μαζί, σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, θέλουμε να διερευνήσουμε την αμυντική διάσταση εκτός από την μη στρατιωτική διάσταση, civil dimension δηλαδή. Θέλουμε κάτι το οποίο να συνεργάζεται αποτελεσματικά. Όμως ο δικός σας κοινοβουλευτικός έλεγχος θα ε, μας βοηθήσει να κλείσουμε όποια κενά ενδεχομένως εντοπιστούν ή αδυναμίες. Απαντώ στην κυρία Μετσόλα για το επιγραμμικό περιεχόμενο, στο οποίο αναφερθήκατε και άλλοι εξημών. Για την ώρα, η συνεργασία που έχουμε, που είναι εθελοντική, πολύ αποδοτική όμως, ιδίω σε ό,τι αφορά το τρομοκρατικό περιεχόμενο σε φόρα του ίντερνετ, έχει σχέση με την αφαίρεση περιεχομένου μετά από γνωστοποίηση, όπως είπατε και εσείς. Το πρόβλημα είναι και κλίμακος και ταχύτητας αφαιρούμε δεκάδες χιλιάδες στοιχεία περιεχομένου, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες. Και τα αφαιρούμε γρήγορα, αλλά όχι αρκετά γρήγορα, διότι πάντοτε έρχεται μερικές ώρες μετά από τη δημοσίευσή του. Εάν μπορέσουμε να είμαστε επιτυχέστεροι σε αυτήν την προσπάθεια, για να γίνει αυτό δηλαδή, χρειαζόμαστε αλλαγή ρυθμού. Και αυτή είναι η πρόκληση την οποία επιβάλλουμε στις εταιρείε και λέμε να συνεργαστούμε για να γίνει αυτόματη η διαδικασία αυτή και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία σας αμέσως ή ενδεχομένως να εμποδίσουμε την ανάρτηση καν του τρομοκρατικού αυτού περιεχομένου. Είναι δύσκολο για πολλούς λόγους. Η κυρία Σαρτζεντίνη με ρώτησε εάν αναθέτουμε εξωτερικά το έργο αυτό σε ιδιωτικούς φορείς ας πούμε. Οι πλατφόρμες υπηρεσιών παίζουν όντως ένα σημαντικό ρόλο, έχουν μια σημαντική ευθύνη εφόσον οι πλατφόρμες τους των ιδιωτικών φορέων χρησιμοποιούνται για την διασπορά του παράνομου υλικού. Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε μαζί τους για να τις βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάχρηση των πλατφορμών τους. Υπάρχει και μια άλλη δύσκολη ερώτηση που έγινε από εσά σχετικά με τον ορισμό του παράνομου περιεχομένου. Υπάρχουν, ε, ε, υπάρχουν όρισμοι συγγνώμη, και στο ερωσιακό δίκαιο και στα εθνικά δίκαια. Και στις χώρες μέλη εφαρμόζονται και τα δύο αυτά και οι δύο αυτοί ορισμοί του παράνομου χαρακτήρα. Χρειάζεται όμως και άλλη συζήτηση σχετικά με την εναρμόνιση της, των προσεγγίσεων εάν σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώνονται διαφορές μεταξύ των ορισμών αυτών. Και Έρχομαι τώρα στην ερώτηση Σπινέλη. Στην προσπάθεια μας αυτή αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να γίνει σεβαστή η ελευθερία έκφρασης και οποιοδήποτε μέτρο προτείνουμε θα είναι απολύτως αναλογικό και αναγκαίο. Αναφέρθηκα και σε μια σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ό,τι αφορά την κλίμακα επενδύσεων στην ασφάλεια. Όχι για θα ήθελα να μεταφέρω άλλες πτυχές του αμερικανικού μοντέλου εδώ, αλλά διότι αυτό που πρέπει να κάνουμε εμεί είναι να φτιάξουμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο, ενωσιακό μοντέλο. Συμφωνώ με την Γεσίπλ για το ότι η συνειδητοποίηση, η ευαισθητοποίηση και η υγιεινή αποτελεί ένα σημαντικό μέρο των προσπαθειών μα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το μικρό έγκλημα, διότι το πρόβλημα με την εγκληματικότητα στο διαδίκτυο είναι ότι πολλές μικρές εγκληματικές πράξεις συναθρίζονται σε μια πάρα πολύ σημαντική πρόκληση. Θα επανέλθω στην κρυπτογράφηση, encryption, γιατί είναι ένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στο πακέτο των προτάσεων CT για την επόμενη εβδομάδα και εκεί θα επανέλθω να σας μιλήσω. Έχουμε όμως προτάσεις για την αντιμετωπίση της κρυπτογράφησης στις ε, ποινικέ έρευνες χωρί ωστόσο να υποσκάψουμε την ακαιρεότητα της κρυπτογράφηση, στην οποία όλοι βασιζόμαστε. Θα τα συζητήσουμε όμω αυτά και με περισσότερε λεπτομέρειε. Τώρα για τα εικονικά νομίσματα. Υπάρχει ορισμός των οικονομικών νομισμάτων στις προτάσεις για πληρωμές, Όμω η Payment Directive, η οδηγία περί πληρωμών, δεν αναφέρεται στην κατάχρηση των εικονικών νομισμάτων για εγκληματικού σκοπού, αναφέρεται στην προστασία κατά απατών σε οποιαδήποτε μορφή πληρωμής, ακόμα και αν χρησιμοποιούνται εικονικές μορφές πληρωμής. Για το ερώτημα της αποτροπής και άμυνας του κ. Ντεπρέ. Ελπίζω ότι έχω ήδη εν μέρει απαντήσει. Για την ώρα οι προσπάθειες κυβερνώ άμυνας είναι κυρίως θέμα των χωρών μελών και εμείς τις στηρίζουμε. Το ζήτημα όμως η έννοια της αποτροπής ξεπερνά την έννοια της άμυνας. Είναι πολύ ευρύτερη, διότι αν το καλοσκεφτείτε, 95, 96, 97, 99% των υπηρεσιών που μπορεί να ε, αντιμετωπίσουν πρόβλημα δεν είναι καθαρά αμυντικά, είναι μη αμυντικού χαρακτήρα, είναι civil. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο ενδεχόμενο επιθέσεων που είναι εκτός του στρατιωτικού αμυντικού τομέα και τα εξετάζουν αυτά άλλες ρυθμιστικές αρχές και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια συνολική προσέγγιση για την αποτροπή για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ένα οπλοστάσιο μέτρων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ε, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις ό,τι αφορά και την ε, προστασία και την ασφάλεια, safety και security, και αυτά θα τα συζητήσουμε όμως σε άλλο πλαίσιο με περισσότερη λεπτομέρεια. Εάν παρέλειψα κάποιες ερωτήσεις σας, ε, να επανέλθετε σας παρακαλώ. Μία σημαντική πρόκληση νομίζω είναι πώς θα προωθήσουμε το έργο αυτό με επιτυχία. Αρχίζει από την Επιτροπή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι συμμετέχουν σε διάφορες πτυχές του έργου πλήρωνες Επίτροποι. Άνσε, Γιουρόβα, Αβραμόπουλος, εγώ προσωπικά και μερικοί άλλοι. Άρα εμεί θα πρέπει να κάνουμε πρώτα σωστά τη δουλειά μα. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό με το σύνολο αυτών προτάσεων που σα υποβάλλουμε. Πρέπει να συνεργαστούμε και με το Συμβούλιο Υπουργών και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ελέγξουμε και να τελειοποιήσουμε τις προτάσεις. Και εκεί χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, γιατί αν δεν μπορέσουμε να συντονιστούμε σωστά, υπάρχει κίνδυνος τελικώς οι προτάσεις να χαθούν μέσα σε μια συνολικότερη συζήτηση και να χάσουμε την ορμή της πρωτοβουλίας. Χρειάζεται όμως να γίνει επίγουσα πρόοδος. Πρόεδρος Μωράης, πριν να φύγετε σε να επανέρχομαι σε κάτι που είπαμε στην αρχή και οι κυρίες Ντάριες και Σπινέλη αναφέρθηκαν στην μεγάλη περιπλοκότητα του χαρτοφυλακίου σας. Θα έρθει μετά να μας μιλήσετε για PNR, για κρυπτογράφηση και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ για την εργασία σας καθώς και ε, την ε, ομάδα σας πάντοτε έχετε προσέλθει όταν σας το έχουμε ζητήσει ενώπιον της Επιτροπής μας έχετε ε, σημαντικούς και ευαίσθητους φακέλους στο χαρτοφυλάκιό σας να συνεχίσουμε την επαφή αυτή έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά από την υπόθεση αυτή της κυβερνοασφάλειας και του κυβερνοεγκρήματος. χρειαζόμαστε πολύ στενή συνεργασία και επαφή με τους πολλούς εμπλεκόμενους επιτρόπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας δούμε την επόμενη εβδομάδα για ακόμα δυσκολότερα θέματα. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις. Ήταν μια πραγματικά πολύ σφιχτή συνεδρίαση. Δεν είμαστε και η μόνη επιτροπή ενώπιον σε εμφανιστήκατε. Έχετε λοιπόν πολύ δουλειά. Πήγατε και στην Επιτροπή του Αγώνα κατά της Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Colleagues, we can move straight to the, our final debate, uh, point 11, this afternoon. Συνάδελφοι, θα περάσουμε κατευθείαν στη τελευταία μας And our commission colleagues will come to the front. I'll start to introduce the item. We have the state of play on the execution of the... Κατάσταση πρόοδο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 στον τομέα μετανάστευσης και εσωτερικών. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που ήρθαν για αυτό το σημείο. And we have the presentation again. Thank you, Simon, for being here. By Simon Mordew, Deputy Director General of DG Home. Colleagues, if you're staying for this item, please. Παρακαλώ, συνάδελφοι, εάν Ε, θέλετε να μείνετε, παρακαλώ να μείνετε ήσυχα. Ο Σάιμον Μόρντιου είναι γενικός αναπληρωτής, μάλλον ε, τη μετάρρηση στη διαθέση TG Home. Και θα μας μιλήσει για την κατάσταση προόδου στην εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2017. Έχουμε λοιπόν την έκθεση της DG Home ως κομμάτι της διαδικασίας για την απαλλαγή για τον προπολογισμό του 2016. Αν το παρακολουθείτε αυτό σημαίνει και το που βρίσκεται η εκτέλεση του προπολογισμού του 2017. Αυτό είναι κομμάτι του ελέγχου που ασκούμε εμείς στο τμήμα 3 του PDP καθώς και το διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 5 επί του προϋπολογισμού του 2017. Όσον αφορά δηλαδή τα 275.000 ευρώ που μεταφέρθηκαν στο νέο Ταμείο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Σάιμον να μας το παρουσιάσετε και μετά θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Ο Σάιμον Μόρτιου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Προσπάθω να συγκεντρώσω όλα τα κομμάτια για να έχετε μια ανέστηση του τι έγινε το 2016, ενώ ταυτόχρονα θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να σας ενημερώσω ε, όχι για το τι έγινε πριν από 9-10 μήνες, αλλά και για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ορισμένε από αυτές, αυτούς τους τομείς κλειδιά, καθώς και για το πού βρισκόμαστε με την εφαρμογή του προπολογισμού και ίσως και ένα-δυο στατιστικές που θα δείχνουν τον αντίκτυπο των όσων κάνουμε μαζί μιλήσω για θέματα που δεν ανέφερε ο Τζούλιαν ή δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Να πω ότι το 2016 ήταν μια αρκετά απαιτητική ε, χρονιά για την DG Home, όπως ξέρετε σε αυτήν την Επιτροπή καλύτερα από όλους, αλλά μπορούμε από την άλλη πλευρά να πούμε ότι έχουν επιτευχθεί απτά αποτελέσματα στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας και προσπαθούμε και να εφαρμόσουμε το συνολικό μας πρόγραμμα για τη μετανάστευση που εκτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη μετανάστευση και θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τους, τις επικεφαλίδες για αυτές τις, ε, αυτές τις ατζέντα, δηλαδή μείωση μετανάστευσης, προστασία εξωτερικών συνόρων, προστασία των όσων το έχουν ανάγκη, καθώς και ε, τακτικά, ε, διαδρομές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστροφή των όσων δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν και τι πρόοδο βρίσκουμε να έχει γίνει ε, στο τομέα των νόμιμων οδών μετανάστευσης για αυτούς που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πολέμηση, κατά της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης, του οργανωμένου εγκλήματος ε, και ε, εμπόριο ανθρώπων, έγκλημα. και πρέπει να πω ότι η άφηξη του Τζούλιαν μας έδωσε μεγάλη πολιτική ορατότητα και έπρεπε να λειτουργήσουμε πολύ πιο εντατικά για να ανταποκριθούμε στις ε, πολιτικές πρωτοβουλίες που εκείνος ανέλαβε. Τι έκαναμε το 2016. Να σας δώσω ένα νούμερο. Είδαμε δραματική αύξηση στη δημοσιονομική ευθύνη και τα κονδύλια της DigiHome. Το 2015 είχαμε 1,7 δις ευρώ. Το 2016 αυτός ο αριθμός σχεδόν διπλασιάστηκε. Από το 1,7 ανήλθε στο 3,2 δις το 2016. Επίσης, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και θα το δείτε από την ετήσια έκθεση διαστηριοτήτων, προσπαθήσαμε να έχουμε σαφείς δείκτες απόδοσης που αξίζει να τους εξετάσει κανείς, αν δεν μπορόλαβε ήδη να το κάνει. Ε, για, εάν επικοινωνείτε με τους ε, εκλογείς σας, έχετε πολλά στοιχεία για το τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα προσπαθήσω κάποια από αυτά τα στοιχεία να τα περιλάβω στην σημερινή μου παρουσίαση. Θα μπορούσα να σας στείλω και ένα-δυο σελίδες ε, που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε στην επαφή σας με τους ψηφοφόρους σας. Τι κάναμε λοιπόν το 2016, να σας δώσω και μια γεύση για το 2017. για την παράνομη μετανάστευση πολύ σαφώς είδαμε τον αριθμό των, να μειώνεται ο αριθμός των παράνομων αφήξεων το 2016 χάρη στη δουλειά μας και τη στενή συνεργασία με τρίτες χώρες καθώς και με τις πρωτοβουλίες που στόχο είχαν να ε, αναχαιτήσουμε τους ε, ε, λαθρέμπορους. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είχε μεγάλο αντίκτυπο στη μείωση των αφήξεων Μάλιστα το 2013-2014 είχαμε ακόμα και 13.000 αφήξεις την ημέρα και στην Τουρκία φτάσαμε, στη συμφωνία με την Τουρκία φτάσαμε στις 80 αφήξεις ημερησίως και κυρίως μειώθηκε η απώλεια ζωών. Εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε με άλλες τρίτες χώρες τώρα. Το 2017 προηγουμένως συζητήσαμε τη δουλειά με τη Λιβύη, με τη, με την Ισία, με χώρες ε, ε, και συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους συναδέλφους στην ΕΙΕΔ. 2016 τονίστηκε περισσότερο η επιστροφή των όσων δεν έχουν δικαίωμα να μείνουν στην Ένωση και που δεν εγκρίθηκε η αιτήσει ασύλου τους. Είχαμε εις βάθος συζήτηση από αυτού πρόσφατα και συμφωνήσαμε να επανέλθω με περισσότερες λεπτομέρειες και για περαιτέρω συζήτηση εντός ολίγου. Αυτό στηρίζεται και από χρηματοδότηση προς τα κράτη-μέλη. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2016 τα κράτη-μέλη δαπάνησαν περίπου 106 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα των επιστροφών. Συνεχίζεται αυτό το 2017. Τονίζω, ενώ σεβόμαστε τις θεμελιώδεις ελευθερίες και όπως ήδη θα είδατε ίσως στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση, οι ιδέες μας τονίζουν τη σημασία του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής που είναι ας πούμε το επιχειρησιακό σκέλος της πολιτικής επιστροφών. Εξακολουθούμε να είμαστε πεπισμένοι πως οι επιστροφές είναι στιγματικό στοιχείο ώστε να υπάρχει αποτροπή ώστε να ξεκινούν οι παράνομες διαδρομές προς την Ένωση, ειδικά για αυτούς που δεν έχουν δικαίωμα σε ε, προστασία ασύλου. Έχουμε 11 ε, αξιωματούχους επαφής στη Σερβία, στη Τινησία, στον Νίγηρα και αλλού. Εργάζονται στις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες στις τρίτες αυτές χώρες και επίσης στη Europol έχει φτιαχτεί ένα ευρωπαϊκό κέντρο για την παράνομη μετανάστευση και μάλιστα είχαμε, έχουμε εκεί συνεργασία ανάμεσα στον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής, της Europol, ώστε να έχουμε ένα συγκεκριμένο κέντρο, ένα κόμβο για να παρακολουθούνται αυτοί οι παράνομοι τόσο εντός Ένωσης όσο και στις τρίτες χώρες. Για τη διαχείριση των συνόρων να τονίσω τη συμβολή της επιχείρησης Τρίτονας και Ποσειδώνας το 2016 αυτές οι επιχειρήσεις επεκτάθηκαν στην Μεσόγειο, να σας δώσω ένα νούμερο, ο αριθμός ζωών που διασώθηκαν στην Κεντρική ε, Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο, χάρη σε αυτές τις επιχειρήσεις, έχουμε 620.000 ζωές που σώθηκαν. Πολύ συγκεκριμένη και θετική συμβολή. Για να συνδεθούμε και με τον προπολογισμό, εδώ λοιπόν δώσαμε και 76 εκατομμύρια ευρώ επίγουσα βοήθεια υπό το ISF για να στηρίξουμε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σημαντικό νούμερο σε δύσκολη ε, αυτή περίοδο με διάφορες πιέσεις που δεχτήκαμε. Ο κανονισμός για τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ήταν από τα πιο σημαντικά που επιτεύθηκαν. Το συζητήσαμε επανελειμμένα, αλλά πούμε ότι ο οργανισμός φτιάχνει τις δυνατότητές της ώστε να παίξει κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Έχουν γίνει αξιολογήσεις, δοκιμές και για τα ευφύ σύνορα και πάλι είδαμε πολύ σημαντική πρόοδο Στη νομοθετική διαδικασία έχουμε πολιτική ε, βούληση και από την δική μας πλευρά έχουμε προτάσεις που ελπίζουμε πως θα έχουν συμφωνηθεί μέχρι τα τέλη του 2017. Hot ε, Έχουμε το σενάριο ανάπτυξης των hotspot με συγκεκριμένες διαδικασίες στάνταρ που επιτρέπουν σε όλες τις υπηρεσίες από την πρώτη άφηξη, την πρώτη γραμμή ψυχολογική στήριξη, ε, πρόσβαση σε νομικές συμβουλές, έλεγχη ασφαλείας έχουν φτιαχτεί και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε να, στηρίξουμε τα κράτη-μέλη που περισσότερο έχουν επηρεαστεί, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η ε, ε, μετανάστες και οι πρόσφυγες καταγράφονται σωστά, ακολουθούνται σκληρές μάλιστα διαδικασίες και ο έλεγχος, ο σκληρός του ελεγκτικού συνεδρίου έδειξε πως λειτουργεί το σύστημα το hotspot και βοηθά στη διαχείριση των μεταναστών, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Μάλιστα τον Οκτώβριο έχουμε πιο λεπτομερείς κατευθυντήριε γραμμές για τις, για τις διαδικασίες στα hot spots. Να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να πω ότι τρία κρατημέλη αντιμετωπίζουν την πιο επίγουσα πίεση στα εξωτερικά του σύνορα και στηρίχτηκαν το 2016 με 210 εκατομμύρια ευρώ επίγουσα βοήθεια από το ISF, η Βουλγαρία 130, 40 η Ελλάδα και 40 η Ιταλία. Το 2016 επίσης ξεκινάμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδο στην ταχύτητα των διαπραγματεύσεων. Το αναφέραμε και στον εκκοινοθέν μας ότι δηλαδή ίσως τα κράτη να μπορέσουν να επιτρέψουν να προχωρήσει αυτή η πρόταση αλλά είμαι πεπισμένος προσωπικά ότι ο, ο, κανονισμός του Δουβλίνου και τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου είναι κρίσιμα για να μπορέσει το σύστημα μας να λειτουργήσει. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα έχουμε διαρκώς καταστάσεις όπου ένα-δύο κράτη αντιμετωπίζουν ε, την μόνιμη, μόνιμα πίεση αδίκως και θα χρειάζονται περισσότερη στήριξη. Επίσης το 2016 έγινε μεγαλύτερη πρόοδος στις μετεγκαταστάσεις. Τα τελευταία στοιχεία στα τέλη του Σεπτεμβρίου Έχουμε φτάσει στις 9.000 μετακαταστάσεις από την Ιταλία και 20.000 από την Ελλάδα. Στην προηγούμενη σύνοδο νομίζω και στον Επίτροπο ρωτήσατε πώς βλέπουμε να συνεχίζονται οι μετακαταστάσεις και η επιλεξιμότητα στην Ελλάδα. Εγώ δεν θα το ανοίξω αυτό το θέμα, αλλά στις δικές μας προβλέψεις για τον προπολογισμό έχουμε διαθέσει χρηματοδότηση ένα δις διατίθεται για στήριξη των προγραμμάτων μετακατάστασης για την ε, με την κατάσταση, δυνατότητα με την κατάσταση σε υπηκόων τρίτων χωρών που χρειάζεται να μετεγκατασταθούν, να ανοίξουμε ένα νόμιμο δρόμο ε, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν διακινητές χωρίς να κινδυνεύσουν και αυτό δείχνει την αλληλεγγύη μας προς τις τρίτες χώρες που φιλοξενούν μεγάλους αριθμούς προσφύγων. Τα τέλη λοιπόν του 2015 φτιάξαμε το πρώτο πανευρωπαϊκό σύστημα επανεγκατάστασης και καταφέραμε 23.000 κόσμο να επανεγκαταστήσουμε με μεγάλο αριθμό Συρίων, με τη δήλωση Ένωσης Τουρκίας. Δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το πνεύμα και τώρα ξεκινήσαμε φιλόδοξη προσπάθεια ώστε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για την επανεγκατάσταση, κατάσταση γύρω στις 50.000 ανθρώπων μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2017. με 500.000 ευρώ πρικοδότηση. 500 εκατομμύρια, συγγνώμη, μισό δις. Πολύ καλό για αρχή. Θέλουμε να εστιάσουμε όχι μόνο στους Συρίους από την Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και για την μετεγκατάσταση, από τη, μάλλον επανεγκατάσταση από την Βόρεια Αφρική και την, το κέρα τη Αφρικής. Ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να βάλει τη ζωή του στα χέρια των διακινητών. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με αυτόν τον μηχανισμό επίγουσες μετακίνησης να φύγουν δηλαδή από τη Λιβύη από τον, προς τον Ήγηρα, προς το Τσάντ και να προσφέρουμε επαναγκατάσταση στην ε, Ένωση. Το να προσελκύσουμε ε, εκπαιδευμένους ε, και με υψηλά προσόντα επικόστη των χωρών είναι η μεταρρύθμιση της μπλε κάρτας που προτάθηκε τον Ιούνιο του 2017. Ορισμένοι θα το είδατε και στη μεσοπρόθεσμη έρευνα. Ξεκίνησε η ιδέα με τα πιλωτικά προγράμματα ώστε να φτιαχτούν νόμιμοι ε, δρόμοι για μετανάστευση, ιδιαίτερα για τη Γουινέα, τη Γάμπια και κάποιες ε, βορειοαφρικανικές χώρες. Τώρα, ριζοσπαστικοποίηση, τρομοκρατία, πολλή δουλειά του 2016, Έχουμε εστιαστεί στην καταπολέμηση των μέσων που χρησιμοποιούν για να κάνουν τις επιθέσεις. Είδαμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας εντός της ε, Europol τον Ιανουάριο του 2016 που βοηθά ώστε να βελτιωθεί ε, η ανταλλαγή πληροφοριών περί ασφάλειας ανάμεσα στις διάφορες αρχές των κρατών μελών. Έχουμε την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης ε, είναι σημαντικό ότι έχουμε προβεί σε δράσεις για να βρούμε λεπτομέρειες και ο Τζούλιαν το τόνισε πριν ώστε να αναχαιτήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση επιγραμμικά. Έχουμε κάνει κάποια πρόοδο. Συνεργασία επίσης με τις ε, εταιρείε ίντερνετ ώστε να αφαιρείται το ριζοσπαστικό ε, περιεχόμενο με αυστηρότερους ελέγχους για τις ε, μεγάλες ροές μετρητών, πάγωμα και κατάσταση περιουσιακών στοιχείων. Έχει γίνει πρόοδο σε αυτά τα στοιχεία. Νομίζω τα ωφέλη θα τα νιώσουν και οι πολίτες μας. Έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο ασφάλειας. 11 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησαν τα κράτη-μέλη στην πρόληψη και την καταπολέμηση καταστάσεων κρίσης και για τη δημιουργία μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης για τρομοκρατικές απόπειρες. Σημαντικό επίτευγμα και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να εντοπίσουμε εντό τη Ένωση ε, και ταξιδιώτε υψηλού κινδύνου που παλιότερα περνούσαν απαρατήρητοι από τι ε, αρχέ και για το οργανωμένο έγκλημα, πολύ δουλειά το 2016, κάναμε προτάσεις για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, την νέα πρόταση για ψυχοδραστικές ουσίες, όπου το Συμβούλιο ε, επίσης συμφώνησε να αναθεωρήσει την ε, οδηγία περί όπλων Το 2016 75 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στα κρατη για την καταπολέμηση των ε, ε, εγκλημάτων και για την πρόληψη αυτών να σας πω δύο πράγματα που με εντυπωσίασαν ε, ε, για να καταλάβετε και να έχετε μια αίσθηση του τι έχει αλλάξει. Αν δείτε το ΣΥΣ, το Σύστημα Πληροφοριών του Σέγγεν, τα στοιχεία του Σέγγεν το 2016 τα συμβουλεύτηκαν τα κράτη-μέλη 3,9 δις φορές ε, ζήτησαν, ζητήθηκαν συμβουλές από το ΣΥΣ. Επίσης είδαμε σημαντική αύξηση στα χτυπήματα σε αυτές τις ε, ε, αναζητήσεις από άποψη είναι σημαντικό αυτό γιατί δείχνει την προστιθέμενη αξία των όσων κάνουμε εδώ, ιδιαίτερα εσεί που φτιάχνετε το νομοθετικό πλαίσιο για όλα αυτά και τον αντίκτυπο των όσων κάνουμε. Σύντομα να σας δώσω μια αίσθηση για το πώς εγώ θα περιέγραφα το πώς παρακολουθούμε τον έλεγχο και τις απαιτήσει ελέγχου, πολύ πίεση και εδώ. Αν δούμε τα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου, κατέληξαν ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου λειτουργούν ικανοποιητικά. Είχαμε θετικά συμπεράσματα το 2015 για συγκεκριμένους ελέγχους για την έμεση, ε, άμεση μάλλον ε, ε, διαχείριση και το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι οι εκτιμήσεις της Κομισιόν επιβεβαιώνονται. Είπαν ότι η Κομισιόν εποπτεύει αποτελεσματικά την εποπτεία των κρατών μελών. Σας εξήγησα και τις διάφορες πρωτοβουλίες. Και έχουμε κάποιους βασικούς ε, δείκτες πάρα πολύ εντυπωσιακού ιδίω. Η αύξηση των ε, πόρων δεν ταιριάζει με τους ανθρώπινους πόρους που δεν γνώρισαν αύξηση. Μεγάλη πίεση υπάρχει επομένως όλοι έχουμε στην υπηρεσία κάθε μέρα και αυτό μια που είμαι υψηλό βαθμός manager με ανησυχεί είναι κακό αυτό για το προσωπικό μας Όσον αφορά την εκτέλεση της χρήσης 2017, πρέπει να σας πω ότι οι επιδόσεις μας είναι σύμφωνες με τις προβολές, αλλά σε δύο τομείς δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Πρώτα-πρώτα η τροποποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου δεν το έχουμε ακόμα αλλά τώρα προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει με τις μετακαταστάσεις να προγραμματιστούμε ούτω ώστε να πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα να πάνε σε αυτούς που τα χρειάζονται και ε, επίση δεν τα πήγαν πάρα καλά με το admission scheme όσον αφορά δηλαδή τις ε, ε, τις υποδοχές όσον αφορά κάποια ε, ε, διαδικασία εθελοντικής ε, συμμετοχής. Όμως θα δούμε τώρα πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις πιστώσεις που έχουμε μέχρι πάντως το τέλος της χρονιάς θα έχει γίνει απορρόφηση όλων των πιστώσεων δείκτης κατανάλωση τέλους Σεπτεμβρίου. Είμαστε στο 72% σε αυτή την ανάλυση των Τρία δις ήταν η πρικοδότηση, άρα 2,2 δις ήδη έχουμε απορροφήσει και αναλώσει. Τα είπαμε για τη μετεγκατάσταση, μην ξαναπώ τα ίδια. Καλά, να βάλω τώρα μια ε, τελεία, αλλά ελπίζω ότι αυτοί οι δείκτες που σας ανέφερα σας κατέδειξαν το ότι κάνουμε τη διαφορά με τη δουλειά μας και ο προϋπολογισμός όντως μας βοηθάει σε αυτή το τόσο, το, τόσο δύσκολο θεματολόγιο πολιτικής που έχουμε. Ευχαριστούμε Σάιμον, μας τα είπες όπως πάντα με πολλές λεπτομέρειες, ε, με μεγάλη πληρότητα και έχουμε την έκθεση του 2016 ε, τώρα είναι το δύσκολο θέμα μετά στο τέλος μιας πολύ δύσκολης μέρας. Ακούσαμε τι γίνεται με όλες αυτές τις ε, πολιτικές. Πάρα πολύ ζώρικα είναι αυτά. Σουρεαλιστικά σχεδόν. Κύριε Μετζόλη, πώ θέλει το λόγο που κάνει νόημα αρνητικό. Όχι. Θέλετε το λόγο, θέλετε. Α, ναι, ναι. να. Μιλήστε, μιλήστε. Κλόντ, σε ευχαριστώ. Εγώ θέλω να μιλήσω σε ένα, για ένα συγκεκριμένο θέμα. Αν θυμάμαι καλά, μας είπατε 106 εκατομμύρια ευρώ για αυτό που θέλω να σας μιλήσω. Τα λέω και τα ξαναλέω σήμερα. Τα ίδια σε όλους μας τους προσκεκλημένους. Αν κάνουμε μια προβολή και κοιτάξουμε τι... Να δούμε. Ποιο είναι το μήνυμα το πολιτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τις επιστροφές, της τους επαναπατρισμούς, τα και στον κύριο Αβραμόπουλο. Αν θέλουμε να έχουμε αξιοπιστία, θα πρέπει να τα πάμε καλύτερα σε αυτό το μέτωπο. Τα 106 εκατομμύρια διατέθησαν. Αν αναλώθηκαν, αν αναλώθηκαν, πώς αναλώθηκαν, γιατί το Συμβούλιο τα λέει και τα ξαναλέει ότι οι συμφωνίες επαρενής θα πρέπει να βελτιωθούν ε, διαπραγματεύσεις με τόσες χώρες, ε, χιλιάδες δηλώσεων, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο να πάμε πέρα από το 36% που έχουμε σήμερα, ε, η αύξηση από το 14% και το 15%. Μα αυτό όμως είναι επειδή βάζουν μαζί και τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλιώς πέφτουν στο 27%. Άρα, τι θα γίνει. Δεν φαινόμαστε και τόσο αποτελεσματικοί σε αυτό το μέτωπο. Άλλες ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Από τον 7 δις που είπατε για κάποια αύξηση προς τα 3 εκατομμύρια σχεδόν αυτό σε σχέση με άλλους τομείς πώς σας φαίνεται αυτή η αύξηση πώς θα μπορούσε κανείς να κατανείμει αυτό το ποσό γιατί η αύξηση είναι τερατώδες για ένα χρόνο για μία χρήση μπορείτε σύντομα να μας δώσετε μια εικόνα του τοπίου έχουμε την ανθρωπιστική βοήθεια Εκεί έχουμε αυξήσει, έχουμε τη συμφωνία με την Τουρκία, αλλά η αναλογική αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο νόμιζα. Τι λέτε. Έχει κάποιο ερώτηση. Όχι. Και πάλι σας ευχαριστούμε αν θέλετε απαντήσετε σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Για τις επιστροφές Πρόκειται για υποχρεώσεις που θα απορροφηθούν. Για την πρόοδο του 2016 είδα μια βελτίωση του αριθμού προσώπων που έλαβαν αποφάσεις επιστροφής και που επεστράφησαν πραγματικά. 46% νομίζω, λίγο πάνω από 45%. Όταν συζητήσαμε πρόσφατα για τις επιστροφές, μία από ένα από τα πράγματα που σας είπα είναι ότι 46% δεν φαίνεται και πολύ. Και είναι και λιγότερο, διότι μέσα στον αριθμό αυτό έχετε μεγάλο αριθμό επιστροφών από τα Δυτικά Βαλκάνια. Γιατί με την απελευθέρωση των προξενικών θεωρήσεων είναι μεγάλη η πρόκληση να συνεργαστούν οι χώρες αυτές μαζί μας. Γιατί αν δεν συνεργαστούν τότε δεν ισχύει πλέον το η ελευθερία των θεωρήσεων. Για άλλες χώρες όμως τα πράγματα είναι, τα νούμερα είναι δραματικά άσχημα, δηλαδή κάτω 10% για χώρες όπως το Μάλι και άλλες. Χρειάζεται λοιπόν να σοβαρευτούμε και να έχουμε να κάνουμε μια εντονότερη προσπάθεια. Κάποια πρόοδος έχει γίνει σε επιστροφές και επανεισδοχές, και τις τελευταίες εβδομάδες ακόμη καταφέραμε να συμφωνήσουμε με την Γουινέα, σημαντική χώρα για την Ιταλία ιδίω σε ό,τι αφορά τις ελεύσεις σε standard operating procedures για, με τον Μπαγκλαντέσιο επίσης προχωρήσαμε και στη συζήτηση για αντικίνητρα Γκάμπια επίσης η ομάδα μου και ο διευθυντής κ. Μισελ ε, πήγαν τόπου, Αιθιοπία, το, το Σαββατοκύριακο επιτευχθεί συμφωνία. Είναι κάτι το οποίο θα είναι πολύ σκληρή δουλειά, αλλά πρέπει να το περιλάβουμε και μέσα στην προσπάθειά μας για συνεργασία με όλους τους εξωτερικούς εταίρους. Ναι, για την προσπάθεια να δημιουργηθούν νόμιμοι διάβλοι, διότι υπάρχουν τομεί όπου χρειαζόμαστε εξειδικευμένο προσωπικό ή ήμι εξειδικευμένο προσωπικό και είναι ενδιαφέρον για τους ανθρώπους αυτούς. 106 εκατομμύρια ακούγονται σαν να είναι πολλά λεφτά, στην πραγματικότητα είναι πολύ λίγα, διότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κίνητρα για εθελοντική επιστροφή πρέπει εκτός από τις αναγκαστικές επιστροφές να ενισχύσετε και τις εθελοντικές επιστροφές. Και εδώ η χρηματοδότηση αρχίζει να αποδίδει. Ένα πρόσφατο παράδειγμα. Λιβύη. Μέσα στο 2017 με χρηματοδότηση από τον ενωσιακό προϋπολογισμό μπορέσαμε να διευκολύνουμε πάνω από 7.000 εθελοντικές επιστροφές πολιτών από την Λιβύη από τη Λιβύη στις χώρες προέλευσής τους. Είναι η δουλειά που κάνουμε για την μετεγκατάσταση. και για τις ε, επίγουσες εκενώσεις από την Λιβύη προς Νιγηρία και Τσάντ. Δίνουμε χρηματοδότηση για αξιοπρεπή πακέτα επιστροφών. Πρόοδος επιτυγχάνεται και με το Αφγανιστάν και εκεί δίνουμε πακέτα χρηματοδότησης για εθελοντικές επιστροφές. Άλλο παράδειγμα η Ιταλία, όπου έχουμε δώσει σημαντική χρηματοδότηση για να αρχίσουν ένα πρόγραμμα εθελοντικών επιστροφών από την Ιταλία και Πολύ περισσότερα χρήματα θα χρειαστούν όμως αν θέλουμε η προσπάθεια να είναι σοβαρή. Κάτι που θα φανεί πολύ σημαντικό είναι να δούμε και πόσο γρήγορα μπορεί η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή μπορεί να στελεχωθεί γρήγορα, διότι εγώ θεωρώ ότι οι αρχές ασύλου των χωρών μελών όταν εκδίδουν μια αρνητική απόφαση πρέπει ταυτόχρονα να εκδίδουν και απόφαση επιστροφής. Πρέπει να υπάρχουν ωστόσο οι συμφωνίες που θα επιτρέψουν να επιστραφεί το πρόσωπο αυτό. Και το ηλεκτρονικό ε, ταχυδρομείο θα πρέπει να φύγει από την ε, πρωτεύουσα να πάει στην κεντρική αρχή για να λέει ότι ο Ιδού αυτή είναι η απόφαση του συγκεκριμένου πρόσωπου να επιστραφεί. Για να είναι αποτελεσματικό το σύστημα και να ανοίξει και περισσότερος χώρος για αυτούς που χρειάζονται γνήσια προστασία. Για τους προϋπολογισμούς δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τίτλος ή άλλο πρόγραμμα μέσα στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης που να έχει δει τέτοια σημαντική αύξηση σε όλους τους τομείς. Σημαντική λοιπόν αύξηση για τα μεταναστευτικά για να στηρίξουμε προσπάθειες της Ιταλίας, της Ελλάδας να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη σημαντική προσπάθεια που γίνεται και για την ακτοφυλακή συνοριαφυλακή αλλά και για το ζήτημα της ασφάλειας. Είναι πραγματικά μοναδική η προσπάθεια και οφείλω να πω σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση το, της τελέχωσης ήμουν πριν στις εξωτερικές σχέσεις και έχουμε μου έδωσαν πολύ περισσότερα χρήματα για στελέχωση, το οποίο δεν συμβαίνει στον τίτλο 3. Οι συνάδελφοί μου της Οικονομικής Διεύθυνσης λοιπόν δεν έχουν την, την ίδια ε, χρηματοδότηση. Μιλήσατε για στελέχωση και πόρους. Και εδώ θα δούμε και το νομοθετικό έργο, διότι την επόμενη εβδομάδα θα δούμε περισσότερη πίεση και στο δικό μας προσωπικό. Και χαίρομαι ε, για αυτό που είπατε για πόρους, γιατί εδώ μας χρειάζονται επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίω για το έργο των ε, Ευρωβουλευτών, όσοι ασχολούνται κυρίω με του δύσκολου αυτού φακέλου, με τριμερεί διαλόγου κλπ. στον χώρο αυτό δικαιοσύνη και εσωτερικών. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. σα ευχαριστώ για την δουλειά που κάνετε και σε εσά και στην ομάδα σας. Ευχαριστώ για την παρουσίαση σήμερα. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι συνάδελφοι ιδίω για το ότι μείνατε μέχρι τέλους. Ευχαριστώ και το προσωπικό. Θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση μας αύριο στις 9. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάποιες επιτροπές που συναντώνται μία φορά το μήνα. Αύριο λοιπόν ξανά ε, στις 9 και θα ξανασυνδεθούμε την επόμενη εβδομάδα. Αύριο λοιπόν.